Uh, Κυρίε και κύριοι, να ξεκινήσουμε. Έχουμε καθυστερήσει 10 λεπτά. Σας παρακαλώ καθίστε. Κυρία Κασπάρη. Καλό απόγευμα σε όλους. Πρόκειται για μια ακρόαση για την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις, για την αγορά δημοσίων συμβάσεων. Ο τίτλος είναι «Βελτίωση της πρόσβασης της αγοράς δημοσίων συμβάσεων, ευκαιρίες και κίνδυνοι» του νέου μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά αυτό αναφέρεται στην πρωτοβουλία της Κομισιόν που ήδη συζητάτε εδώ στο Κοινοβούλιο. Να ξεκινήσω υπενθυμίζοντάς σας ότι η Κομισιόν υπέβαλε μια πρόταση πέρσι το Μάρτιο για ένα σχετικό μέσο. Αυτή η πρόταση είναι μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να συζητήσουμε. Και αυτό το κοινοβούλιο αρέσκεται στο να συζητά πριν ε, να λαμβάνει αποφάσεις, γι' αυτό θεωρήσαμε ότι χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για το πιθανό αντίκτυπο αυτής της ε, πρωτοβουλίας πριν οι συνομοθέτες να μπορέσουν να προσδιορίσουν τις αντίστοιχες θέσεις τους. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια δημόσια ακρόση για το θέμα αυτό με εμπειρογνώμονες ε, και ειδικού προκειμένου να ρίξουμε περισσότερο φως στα ζητήματα αυτά. Σίγουρα οι εμπειρογνώμονες και τα σχόλιά τους θα συμβάλλουν στις δικές μας συζητήσεις και ο κύριος Κασπάρη που είναι ο εισηγητής και καθίστε στην πρώτη σειρά αυτής της αίθουσας θα μέσα στη σχολιά του Έχουμε δύο πάνελ οργανώσει. Το πρώτο αφορά του κινδύνους και ωφέλη της αμοιβαιότητα στο άνοιγμα των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Σε αυτό το πάνελ έχουμε δύο μιλητέ. Η πρώτη ομιλία θα υλοποιηθεί από τον κύριο Νίκολα Σνίγκλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής προστάμενος του μετός του ΠΟΕ. Ανήκει στην αντιπροσωπεία της Ελβετίας, στον ΠΟΕ. Και ασχολείται με την Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Θα μας μιλήσει για το δίκαιο του ΠΟΕ και τις Δημόσιες Συμβάσεις στο Διεθνές Εμπόριο και ο δεύτερος ομιλητής ε, θα είναι ένα συνήθις προσκεκλημένος αυτή της επιτροπή, ο κύριος Στέφεν Γούλκοκ από το London School of Economics, ο οποίος θα μας μιλήσει για την αξιολόγηση του προτιμονού μέσου, για τη δημιουργία διαπραγματευτικού πλεονεκτήματος, παρουσίαση της μελέτης που ανατέθηκε από την Επιτροπή μας. Τους ορίζω και τους δύο. Να δώσω το λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Νίγκλη. Πού είστε, έχετε το λόγο. Ξέχασα να σας πω ότι έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας, ο καθομιλητής. In order to leave, uh, plenty of... Έτσι ώστε να αφήσουμε αρκετό χρόνο για τη συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να πάρω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ τα μέλη του Κοινοβουλίου, τους αξιότιμους βουλευτές που μου δίνουν τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή την ακρόαση. Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο προκλήσεις που η γραμματεία παρουσίασε σε μας. Μου είπαν ότι πρέπει να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Αν μιλήσω όμως στα γερμανικά, τη διάλεκτο, την ελβετική, καταλαβαίνετε ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβουν τίποτα. Ας αφήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Ξέρω ότι δεν έχουμε προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, μου δίνετε 10 λεπτά. 10 λεπτά για ένα πάρα πάρα πολύ περίπλοκο θέμα και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ακόμα πιο μεγάλη πρόκληση από το να ανοίξουμε όλες τις αγορές δημόσιων προμηθειών στον κόσμο. Θα ξεκινήσω λοιπόν με κάποια σχόλια. Έχω την τιμή και το πλεονέκτημα να συνεργαστώ από το 2010 στο 2012 με το θέμα αυτό στα πλαίσια του ΠΟΕ στην Γενέβη και θα σας μιλήσω εδώ αν θέλετε υπό το πρίσμα αυτών που έγιναν στην Γενέβη. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων και νομίζω αυτό είναι σημαντικό και πρέπει να το πούμε στην αρχή αυτής της παρουσίασης θα πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα έδειξε πάρα πολύ ε, δυναμική θέση όσον αφορά το άνοιγμα των αγορών, τη διαφάνεια, την καλύτερη χρήση των ε, κονδυλίων που προέρχονται από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι ομιλητές συνήθως παρουσιάζουν τρία σημεία στις ομιλίες τους. Εσείς όμως είσαστε πάρα πολύ έξυπνο κοινό. Επιτρέψτε μου λοιπόν να προσθέσω άλλο ένα σημείο σε αυτά τα παραδοσιακά τρία μίας ομιλίας. Καταρχήν, θα σας πω ότι ένας καθαρός, φρέσκος αέρας μας έρχεται από τη Γενέβη. Ναι, Ήδη από το Δεκέμβριο του 2011 είδαμε κάποια αποτελέσματα μετά από 10 χρόνια διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό και σε Υπουργικό Συμβούλιο μπορούμε να πούμε ότι φτάσαμε σε μια συμφωνία. Και πραγματικά τα αποτελέσματα αυτά είναι ιστορικά αποτελέσματα και θα σας εξηγήσω τώρα γιατί. Ίσως όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης, η νέα αυτή συμφωνία θα είναι κατά κάποιο τρόπο σαν την τρίανα του Ποσειδώνα. και κατά κάποιο τρόπο θα αποτελέσει ένα πακέτο κινήτρων γιατί καταφέραμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση να δημιουργήσουμε νέα πρόσβαση στις αγορές για πάνω από εκατοντάδες δισεκατομμύρια το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη θέση της και την διαπραγμάτευσή της. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση όσον αφορά την προηγούμενη συμφωνία του 1995 και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι διατάξεις της νέας συμφωνίας μπορούν να συμπεριλάβουν όλα τα μέλη τα οποία δεν έχουν ακόμα προσχωρήσει στον ΠΟΕ αλλά θα το κάνουν. Και τρίτον, σήμερα έχουμε πρόγραμμα εργασιών για το μέλλον για την αντιμετώπιση θεμάτων όπως παραδείγματος χάρη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι δημόσιες προμήθειες, η διαφάνεια και διάφορα θέματα τα οποία έλειπαν από την προηγούμενη συμφωνία. Γι' αυτό και πάλι θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν είναι διαθέσιμη αυτή η νέα συμφωνία για να ανοίξουν οι αγορές και αυτό το νέο εργαλείο μας επιτρέπει να δούμε ίσως λίγο καλύτερα το τι θα μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και αναβαθμίσαμε αυτήν την συμφωνία που σήμερα έχει γίνει ο ακραγωνιαίος λίθου αυτού του πολυμερού συστήματος για τις εμπορικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε αυτή η συμφωνία πρέπει να σας πω ότι έχουμε δει μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος Πρόκειται, όπως σας είπα, για ένα νέο εργαλείο, για έναν φρέσκο άνεμο, ο οποίος ε, φυσάει από τη Γενέβη προς τον υπόλοιπο κόσμο και αυτό πραγματικά θα δημιουργήσει ένα διαφορετικό περιβάλλον. Γιατί, είναι η πρώτη ερώτηση, γιατί οι χώρες που σήμερα δεν ανήκουν στον ΠΟΕ και δεν ανήκουν και δεν έχουν προσχωρήσει στην συμφωνία, γιατί σήμερα μπορεί να ενδιαφερθούν να γίνουν μέλη. Αυτό πρώτον γιατί αν κάποιος προσχωρήσει σε αυτήν την συμφωνία θα έχει καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, θα έχει προστασία από τον προστατευτισμό και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Πολλές μεταρρυθμίσεις έχουν ε, γίνει σε πολλές χώρες όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες και πολλές φορές μέσω αυτών των ε, μεταρρυθμίσεων που έγιναν χωρίς ε, εξωτερική πίεση οδηγούνται οι χώρες σε καλύτερη διακυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι η διαφορά, η διαφορά και η κακή διακυβέρνηση έχουν ένα πολύ σημαντικό κόστος, αλλά ίσως κάποιος ο οποίος ανήκει ε, στον ΠΟΕ αλλά δεν ανήκει σε αυτήν την συμφωνία, ίσως θα ενδιαφερθεί Δεν ξέρω πόσα είναι τα μέλη ακριβώς αυτή τη στιγμή που έχουν προσχωρήσει, αλλά πραγματικά πάνω από 40, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα και θα πρέπει εδώ να δούμε ακριβώς τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε ένα κίνητρο ή μία τιμωρία. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, ίσως και τα δύο χρειάζονται. Θα σας παρουσιάσω παρόλα αυτά κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνονται αρκετά ενδιαφέροντα για τα οποία θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε. Και θα ξεκινήσω μιλώντας για τον Καναδά και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων Πρέπει να σας πω ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ξεκίνησαν με μια προστατευτική προσέγγιση οχυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την αγορά τους, ε, προστατεύοντα τις από τους Καναδούς και είδαμε ότι η απάντηση των Καναδών ε, τους οδήγησαν τελικά σε μια διαφορετική προσέγγιση και στο άνοιγμα της αγοράς τους όλες οι χώρες θα πρέπει να συμπεριφερθούν έτσι. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ και είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς εκ των υστέρων σε αυτήν την ερώτηση. Η πολιτική διάσταση τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν θέλει να κλείσει τις αγορές της, γιατί πάντα η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αντίθετη προς το κλείσιμο και την προστατευτισμό. Όμως, το θέμα δεν είναι ποια είναι η μέχρι τώρα τάση. Το θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται ο εξωτερικός κόσμος την πολιτική που υιοθετεί μια περιοχή ή ένα κράτος. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ερωτηματικό. Και θα είναι πολύ κρίμα να οδηγηθούμε εδώ σε μια κατάσταση που δεν θα υπάρχουν πλεονεκτήματα για κανέναν. Τώρα, όσον αφορά τους κανόνες, και εδώ η κατάσταση είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Πρέπει να σας πω ότι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και πολύ λίγες απαντήσεις. Αναρωτιάμαστε λοιπόν εδώ από πού προήλθαν οι πρώτοι κανόνες. παραδείγματος χάριν για την αγορά του κρέατος. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να παρακολουθήσουμε, παραδείγματο χάρη, την προέλευση ενός προϊόντος. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά ένα θέμα σε γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν κανόνες, θα πρέπει αυτά που θα υιοθετήσει να είναι μέτρα τα οποία να συμμορφώνονται με τους κανόνες ε, της ε, σύμβασης αυτής και σαν επικεφαλής ε, του, της υπηρεσίας αυτής του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου θα πρέπει να σας το πω. Εδώ πρέπει να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών κανόνων και αυτών του ΠΟΕ. Θα πρέπει επίσης να σας πω ότι εδώ αναφερόμαστε για 30 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και για το 25% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παίζει έναν ηγετικό ρόλο στον τομέα των ε, δημόσιων συμβάσεων, την τελευταία δεκαετία έχει παίξει καθοριστικό ρόλο τροποποιώντας ε, την, το σκηνικό σε διεθνές επίπεδο με πολύ καθοριστικό τρόπο και η νέα αυτή συμφωνία σίγουρα θα οδηγήσει σε πολύ θετικά αποτελέσματα. Είμαι σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση θα κερδίσει, θα επωφεληθεί από αυτό το νέο σκηνικό και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ότι αν δούμε διαφορετικές συμπεριφορές όπως αυτή που είδαμε παραδείγματος χάρη από τις Ηνωμένε Πολιτείες το 2008-2009 αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να έχει αποτελέσματα εκτός αυτού του πλαισίου των συμφωνιών. Έχω λοιπόν εμπιστοσύνη όσον αφορά την εξέλιξη ε, αυτής της συμφωνίας. Σας ε, έθεσα σίγουρα πολλά ερωτήματα, πολύ περισσότερα από τις απαντήσεις που σας έδωσα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι προοπτικές αυτές που μπορούμε σήμερα να δούμε και να σχεδιάσουμε από τη Γενέβη είναι σίγουρα πολύ καλύτερες από αυτές του παρελθόντος και ελπίζω να ήμουν χρήσιμος με την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής ο κύριος Στέφεν Γουλκοκ ε, ε, από το London School of Economics, όπως σας ενημέρωσα ήδη, θα μας παρουσιάσει τη μελέτη που ζητήθηκε από αυτή την Επιτροπή, από το London School of Economics, ε, από την Μονάδα Πολιτικής Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μείνω στα 10 λεπτά. Πρόεδρε, της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στα 10 λεπτά θα προσπαθήσω να συνοψίσω τη μελέτη. Όπως ε, είπε και ο κύριος ε, Νίκλε, είναι πολύ πλοκό αυτό το θέμα και περισσότερο αφορά ένα θέμα κρίσης από ότι στα περισσότερα εμπορικά ζητήματα, γιατί υπάρχουν μη επαρκή δεδομένα, αν και η Κομισιόν έχει, κάνει, έχει βάλει τα δυνατά της για να πληρώσει τα κενά και υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σε σχέση με το αν είναι καλό να υιοθετήσει μία πιο σκληρή γραμμή για την αμοιβαιότητα. Επίσης, είναι δύσκολο να κρίνει κανείς το αποτέλεσμα, γιατί πολλά εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιείται στην πράξη ο κανονισμός και πώς θα απαντήσουν οι χώρες. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οντότητες που αγοράζουν τείνουν να ευνοούν την ε, μη ανάληψη δράσης, ε, γιατί μπορεί να είναι πιο πολύπλοκο ε, το εγχείρημα και τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά σε ορισμένους τομείς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από εθνικούς πρωταγωνιστές σε άλλες αγορές. Αυτοί θέλουν να δουν να προχωρήσει ο κανονισμός, όμως γενικά οι επιχειρηματικές ενώσεις έχουν μία πιο μεικτή θέση, κάποιοι είναι υπέρ, κάποιοι είναι κατά. Και αυτό ισχύει για τα κράτη-μέλη. Αυτό που θα κάνω εγώ είναι να αναφερθώ σε τέσσερα ζητήματα. Καταρχήν, το θέμα, το πώς ε, το σχετικός ανοιχτός χαρακτήρας της ε, ε, ευρωπαϊκής αγοράς εναντί άλλων αγορών. Δεύτερον, το κόστος και το όφελος της χρήσης του κανονισμού κατόπιν, αν είναι προστατευτικό ή όχι και αν θα λειτουργήσει. σχέση με την πρώτη ερώτηση, αυτό είναι ένα από τους τομείς όπου δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη. Υπάρχουν ε, μελέτες που λαμβάνουν ε, ε, μια ευρεία εικόνα των δημοσίων συμβάσεων και μετρούν την κατανάλωση. Το πόρισμα αυτών είναι ότι είναι λιγότερο ανοιχτή η ευρωπαϊκή αγορά από ό,τι στην Ινδία και την Κίνα, λίγο πιο ανοιχτή από ό,τι στις Ηνωμένες και λίγο πιο ανοιχτή από ό,τι στην Ιαπωνία. Και αυτό μπορεί να μας εκπλήσει κάπως, όμως ε, αν ε, δούμε ε, τα συνολικά νούμερα, αυτό, αυτό βασίζεται στα συνολικά νούμερα που περιλαμβάνουν όλους τους τομείς, την εκπαίδευση, τα πάντα. Αν ε, κάνουμε κάποια επιμέρους ανάλυση και δούμε επιμέρους τομείς, έχουμε πολύ διαφορετική εικόνα και αυτό ακριβώς έκανε η Κομισιόν στη μελέτη αντικτύπου. Αν δούμε βασικούς τομείς ε, που φαίνεται να είναι στρατηγικής ε, σημασίας, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η άμυνα, μεταφορές, ιατρικός εξοπλισμός, οι κατασκευές, η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι πιο ανοιχτή η ευρωπαϊκή αγορά σε σχέση με άλλες αγορές. Υπάρχουν ε, βέβαια και άλλες πτυχές σε αυτό και συγκεκριμένα η πρόσβαση στις ε, δημόσιες ε, συμβάσεις γίνεται πιο συχνά μέσω μιας τοπικής θηγατρικής ή ενός τοπικού υποκαταστήματος. Αν ε, δείτε την πρόσβαση στις ε, αγορές δημοσίου συμβάσεων των κρατών μελών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, θα δείτε ότι περίπου το 4% των μη κρατών μελών αντιστοιχεί στο 14% που κάνουν έτσι, αντιστοιχεί στο 14% των συμβάσεων και αυτό γίνεται κυρίως μέσω θυγατρικών και κυρίως προέλευσης ΩΣΑ. Έτσι λοιπόν θα περίμενε κανείς ε, ε, εκεί να συναντήσει τις Ηνωμένε Πολιτείε, την Ελβετία και άλλους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά προσφέρει διαφάνεια στις δημόσιες ε, συμβάσεις. Επίσης, είναι ένα φιλελεύθερο καθεστώς για τις επενδύσεις, έτσι λοιπόν θέλει κανείς να έχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω ενός υποκαταστήματος, αυτό είναι σχετικά εύκολο. Και η διάκριση που γίνεται στη συζήτηση σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις μεταξύ διαφάνειας και απελευθέρωσης, νομίζω πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά. Αν έχει κανείς διαφάνεια, αυτό σημαίνει ότι ανοίγει και η αγορά στον ανταγωνισμό. Και τέλος, για αυτό το θέμα, οι μεγάλες αναπτυγμένες ε, οικονομίες που βασίζονται στην αγορά συνηθίζουν να έχουν λιγότερες εισαγωγές από οι λιγότερο αναπτυγμένες αγορές γιατί έχουν ικανότητα εγχώριας προμήθειας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προμηθεύει και να καλύπτει τη μεγαλύτερη αποτιζήτηση από εσωτερικούς προμηθευτές. Δεν χρειάζεται να βασίζεται και να αντιλήξαν ανταγωνισμό αυτό σχετίζεται με τη συζήτηση γιατί πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ε, είναι διστακτικές να δεσμευτούν σε θέματα δημοσίων συμβάσεων. Έτσι λοιπόν, ε, κάποιο πρέπει να κάνει μια κρίση εδώ, γιατί δεν υπάρχουν ξεκαθαρά αριθμητικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι το συμπέρασμα είναι μπορεί η ευρωπαϊκή αγορά να είναι πιο ανοιχτή σε ορισμένου τομεί, αλλά αν έχουμε μια πιο γενική εικόνα, βλέπουμε ότι δεν είναι πιο ανοιχτή από τη άλλη να προχωρήσουμε τώρα στο πιθανό κόστος ε, και στα ωφέλη και πάλι οι δυσκολίες εδώ είναι ότι έχει γίνει πολύ λίγη δουλειά στον οικονομικό κόσμο σε σχέση με το γενικό κόστος και τα ωφέλη των καθεστώτων συμβάσεων. Είναι πολύ πιο εύκολο να εργαστεί κανείς ε, για τους δασμούς, ε, ακόμη και για τους μη δασμολογικούς εφραγμούς, είναι πιο εύκολο να αξιολογηθεί αυτό, αλλά είναι δύσκολο να αξιολογηθεί το κόστος και το όφελος του ανοίγματο ε, των αγορών δημοσίων συμβάσεων. Η Κομισιόν στη μελέτη αντικτύπου λέει ότι τα ωφέλη θα προκύψουν από αυξανόμενε εξαγωγέ και από αυξανόμενε από εργασία θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα σε ορισμένου στοχευμένου τομεί. Αυτή είναι η τομείς όπου οι διεθνείς ε, πρωταγωνιστές ε, τρίτες χώρες έχουν ε, κάποια επιθετικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν έχουν τέτοια επιθετικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε μπορεί να θέλουν να απαντήσουν περισσότερο στην απειλή του κλεισίματος της αγοράς. Επίσης, ε, σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό, θα αυξηθεί η μόχλευση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις, η διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην ευρωπαϊκή πολιτική μέσω του κανονισμού, γιατί αυτή τη στιγμή με τι υφιστάμενε διατάξεις, συγκεκριμένα τον κανονισμό 17 του 2004, για οι οντότητες, οι μεμονωμένες οντότητες που αγοράζουν μπορούν ε, να εφαρμόσουν μέτρα αμοιβαιότητα κατά συγκεκριμένων χωρών και αν το κάνουν αυτό, αυτό θα υποβαθμίσει, θα υποσκάψει την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος, έχετε αυτό το γενικό ερώτημα για το πιο γενικό θέμα για λιγότερο αποτελεσματική χρήση των δημοσίων δαπανών. Δεν υπάρχουν εδώ κατάλληλα αριθμητικά στοιχεία. Επίσης υπάρχει το κόστος ε, της συμμόρφωσης που ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουμένω ε, σε σχέση με τους κανόνες προέλευση, ιδίω, αλλά οι οντότητε ε, θα αντιμετωπίσουν μεγάλο κόστος για τη συμμόρφωση, αν και η Κομισιόν δεν πιστεύει κάτι τέτοιο στη μελέτη αντικτύπου. Υπάρχει και το πιθανό, η πιθανότητα αντιποθετικών μέτρων κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπάρχει και ζημιά στην εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ε, φιλελεύθερο εμπορευμένου και σε αυτό αναφέρθηκε ο κ. Νίκλο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει για το άνοιγμα των δημοσίων ε, συμβάσεων για λόγους ε, καλής διακυβέρνησης και αποτελεσματικής χρήσης των δημοσιονομικών, των δημοσίων πόρων. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι εδώ η κρίση πρέπει να είναι η εξής. Οι πληροφορίες απλώς δεν είναι διαθέσιμες για να προβούμε σε μια σωστή αξιολόγηση κόστους και ωφέλους και εξαρτάται από το πώς θα χρησιμοποιηθεί ο κανονισμός. Μου τελειώνει ο χρόνος, Πρόεδρε. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα όμως δεν μπορεί να κρυθεί αυτό το θέμα. Είναι πολύ υποκειμενικό, αλλά αυτό που μπορούμε να κρίνουμε είναι ότι ο βαθμός της αμοιβαιότητας αν ορίζεται στενότερα στενότερη ευρωπαϊκή πολιτική ορίζει γενικά την αμοιβαιότητα με ευρύ όρους, ευρέως, δηλαδή στην ορολογία του ΠΟΕ χρησιμοποιούμε παγκόσμια αμοιβαιότητα. Το νερό αυτό, αν υιοθετηθεί ο κανονισμός, νομίζω ότι θα θεωρηθεί ως μετάβαση προς τη στενή αμοιβαιότητα. Και τέλος, σε σχέση με το αν αυτό θα λειτουργήσει, μπορώ να πω κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Το άνοιγμα των δημοσίων συμβάσεων ε, δεν ε, θα επιτευχθεί μόνο με τη σύναψη μια συμφωνία, ακόμη και αν πρόκειται για συμφωνία δημοσίων συμβάσεων ή για μια προτιμεσιακή εμπορική συμφωνία. Υπάρχουν πολλά κρυφά μέσα με τα οποία μπορεί να κρατήσει κανείς κλειστές τις αγορές του. Και υπάρχει αυτό σε όλες τις ε, αγορές δημοσίων συμβάσεων. Έτσι λοιπόν το να πούμε ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούμε ε, προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες ε, και συμφωνίες περί δημοσίου συμβάσεων είναι μια καλή στρατηγική, αλλά αυτό μπορεί να μην αρκεί σε τομείς όπου έχουμε εθνικούς πρωταγωνιστές ε, που προσπαθούν να ανταγωνιστούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Και κάποιος θα μπορούσε να πει επομένω ότι η πολύ περιορισμένη χρήση της εμβεβαιότητας μπορεί να έχει κάποιο όφελος. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γούλκοκ. Ας περάσουμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Οι εμπειρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετοχές σε αγορές δημοσίων συμβάσεων. Τώρα έχουμε πάλι δύο μιλητές. Ο πρώτος ε, προέρχεται από τη Γερμανία, ο κύριος Χάικο Χάινρις. Ευκαιρίες και προκλήσεις με τη συμμετοχή τρίτων χωρών σε δημοσίους διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, δυνατότητα υλοποίηση του προτινόμενου μέσου. Παρακαλώ, που είστε. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, ήθελα να σας ευχαριστήσω εγκάρδια για την πρόσκληση σε αυτή την ακρόαση. Να σας πω δύο λόγια για μένα. Ονομάζομαι Χάικο Χάινριξ. Είμαι υπεύθυνο τη Κεντρική Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων, μια τοπική αναθέτουσα αρχή του Rhein Neuss στη Γερμανία. Και εκεί είμαι υπεύθυνο για την διαξαγωγή ε, αναθέσεων έργων και για την υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών όσον αφορά τι νομικέ απόψει των συμβάσεων. Με αυτή την αρμοδιότητα θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τις ε, δικές μου εκτιμήσεις ως ε, υπαλλήλου σε αυτόν τον τομέα που μας έχει δημιουργήσει το πρώτο επίπεδο των διατάξεων. Καταρχάς, χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δημιουργήσει δίκαιους κανόνες για, τους, για την πρόσβαση στην αγορά οικονομικών φορέων τρίτων ε, κοινοτικών οικονομικών φορέων για τις αγορές ε, προμηθειών στις τρίτες χώρες, αλλά και ε, το αντίθετο. Τώρα, εάν το δίκαιο των συμβάσεων και συγκεκριμένα ο κανονισμός αυτός είναι γενικά ο σωστός για να επιτύχει τον πολιτικό σκοπό, ε, θα σας διατυπώσω ακολούθως τις εντυπώσεις μου. Ο κανονισμός αυτός για εμάς ως εντολής δημοσίων συμβάσεων είναι κυρίως, προορίζεται κυρίως ε, για μεγάλα τεχνικά έργα, για τηλεπικοινωνίες, για κέντρα συντονισμού πυροσβεστικών ε, υπηρεσιών, υπηρεσιών διάσωσης ή χρηματοπιστωτικού λογισμικού. Και θα μας ε, χρησιμεύσει λοιπόν για τους τομείς αυτούς καθώς και, αυτούς, καθώς και για μεγάλα έργα υποδομής. Ε, ορισμένα σημεία αυτού του κανονισμού τα βλέπω με κριτική άποψη όσον αφορά τις πρακτικές εφαρμογές τους και την εκτελεσιμότητά τους. Ε, μέσω αυτού του κανονισμού αυτό που βλέπουμε είναι εκτός από τις υποχρεώσεις για συντονισμό των συμβάσεων με επιπλέον υποχρεώσεις ε, εξακρίβωσης. Ε, βλέπουμε λοιπόν πως δημιουργούνται ιδιαίτερα, μεγάλος, ε, ιδιαίτερα μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Και αντίθετα από τον κύριο Νίγκλη θα σας αναφέρω τρία παραδείγματα. Θα περιοριστώ σε τρία. Καταρχάς, πρέπει να υποχρεώσουμε τους υποβάλλοντες προσφορά στα πλαίσια με υπεύθυνε δηλώσεις να πληρούν όλες τις τυπικές ε, προϋποθέσεις του τελωνιακού δικαίου για την ε, προέλευση των αγαθών και των υπηρεσιών τους. Έπειτα, όταν ζητούμε μια ε, έναν αποκλεισμό προσφοράς, ρισκάρουμε να παραταθεί η διαδικασία προσφοράς σε δύο μήνες και πολλές και εάν υπάρξει παράταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παράταση τεσσάρων μηνών. Επίσης, τρίτον, πριν την ανάθεση μιας σύμβασης, πρέπει να εξακριβωθεί εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη λάβει περιοριστικά μέτρα ενάντια σε μια τρίτη χώρα ή σε μια συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών από αυτήν την χώρα. Όλα αυτά κάνουν μια ήδη περίπλοκη ε, διαδικασία ακόμα πιο περίπλοκη και χρονοβόρα. Κυρίε και κύριοι, πρέπει να σκεφτείτε ότι λόγω του μεγάλου αριθμού, ε, του, του μεγάλου όγκου ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, ένα ε, μέσο διοικητικό υπάλληλο όπω εγώ δεν είναι πλέον σε θέση να διεξάγει επιτυχώ μία διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μόνος του και αυτό που έχει οδηγήσει, αυτό έχει οδηγήσει ε, εμάς τους αναθέτοντες φορείς να προσλάβουμε εμπειρογνώμονες και νομικούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στο δίκαιο αυτό των δημοσίων συμβάσεων και αυτό ανεβάζει φυσικά το κόστος πάρα πολύ. Επίσης, να επιθυμίσω ότι ο, κόστος, ότι ο στόχος είναι η απαλλαγή από την γραφειοκρατία. Όμως, ο κανονισμός αυτός, έτσι όπως έχει συσταθεί, οδηγεί σε ακόμα περισσότερη γραφειοκρατία και νομική ασάφεια. Ο δικός μας στόχος, ως αναθέτουσες αρχές, είναι καταρχάς να καλύψουμε τις οικονομικές ανάγκες, ε, με, λαμβάνοντας υπόψη την τιμή και την ποιότητα. Επίσης, ε, σε αυτό, το, σε αυτό το σημείο βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, απόψεις οι οποίες δεν έχουν ε, να κάνουν απόλυτη σχέση με το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, αλλά με δευτερογενεί τομεί, όπως για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος, την καινοτομία, κοινωνικές απόψει και τι διεθνεί εμπορικέ σχέσει. Επίσης, οι κανονισμοί, όπως σας είπα, γίνονται ακόμα περισσότερο περίπλοκοι. Και ως αποτέλεσμα όλων ε, αυτών μου δημιουργείται το ερώτημα εάν θα υπάρξει ε, το ενδιαφέρον εάν μάλλον, σε περίπτωση μάλλον που ζητηθεί ε, αποκλεισμός προσφοράς, εάν αυτό θα μπορέσει να ε, δρομολογηθεί. Στην περίπτωση αυτή, σε μια περίπτωση αποκλεισμού προσφοράς δηλαδή, πρέπει να ε, εξετάσουμε και να εξακριβώσουμε εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ε, λάβει, όπως σας είπα, περιοριστικά μέτρα. Τώρα, όσον αφορά τη διάρκεια της διαδικασίας συμβάσεων. Στην περίπτωση όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάσει τον πιθανό αποκλεισμό μιας προσφοράς, τότε παρατείνεται η διαδικασία ε, των ε, προσφορών για τις δημόσιες συμβάσεις και των διαγωνισμών. Αυτή η προθεσμία μπορεί να διαρκέσει από δύο έως τέσσερις μήνες. Και αυτό ε, δεν είναι δεν είναι εφικτό στα πλαίσια μιας ε, διαδικασίας τέτοιας ε, σύμβασης. Επίσης, μια τυπική τέτοια διαδικασία για συντονισμό συμβάσεων διαρκεί 7 εβδομάδες από τη δημοσίευση της, ε, του διαγωνισμού μέχρι την υποβολή προσφοράς. Και με τον κανονισμό αυτό ενδέχεται να, επεκταθεί, να παραταθεί μάλλον η, το χρονικό πλαίσιο σε τρεις μήνες. Και σε περίπτωση που μια τρίτη χώρα διαπιστωθεί ότι παρουσιάζονται περιορισμοί όσον αφορά τους, ε, τους, ε, του φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρονται, η διαδικασία αυτή μπορεί να παρατεθεί μέχρι και τους πέντε μήνες. Και ο σκοπός της διαδικασία μιας ε, ανάθεσης σε μια σύμβαση είναι η διαδικασία αυτή να ολοκληρωθεί όσο το δυνατόν συντομότερο. Και αυτό με τον παρόν κανονισμό δεν είναι δυνατόν. Τώρα, ε, υπάρχουν προβλήματα με τον χαρακτηρισμό προέλευσης. Ας υποθέσουμε ότι υποβάλλεται ένα, ερώτημα για, ε, ε, ένα αίτημα για αποκλεισμό προσφοράς ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένοι τυπικοί κανόνες. Για παράδειγμα, έχουμε από τον υποβάλλον προσφορά μια υπεύθυνη δήλωση για την προέλευση των, των αγαθών και υπηρεσιών του, και επίση πρέπει να εξακριβώσουμε εάν πληρούνται οι διατάξεις τελωνιακού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 3. Και εδώ έχουμε διαπιστώσει προβλήματα τα οποία επαναλαμβάνονται. Πολλές φορές ε, υποβάλλονται σε προσφορά έχουν ε, ε, υπερβολικά μεγάλο φόρτο διοικητικό όσον αφορά την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων και πολλές φορές οι ίδιοι ούτε, ούτε ξέρουν ούτε και μπορούν να αποδείξουν πλέον την προέλευση των ε, αγαθών και των ε, υπηρεσιών τους. Και αυτό οδηγεί πολλές φορές σε ελλειπή ή ε, λάθος, λανθασμένα στοιχεία. Και αυτό, αυτό το βλέπω κάθε μέρα στην πράξη και εμείς. Και δεν, είναι, δεν συμβαίνει μόνο στους ε, υποβάλλοντες προσφορά, αλλά και σε εμάς ως ε, αναθέτοντες. Ε, πρέπει... Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε με ακρίβεια την προέλευση των αγαθών και των υπηρεσιών μας εάν, εφόσον, εάν μας λείπουν τα μέσα γι' αυτό, το know-how και οι ικανότητες. Πρέπει δηλαδή να εμπιστευόμαστε τις υπεύθυνε δηλώσεις των υποψηφίων χωρίς να μπορούμε αυτό να το εξακριβώσουμε. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να εξακριβώσουμε για ένα κατασκευαστικό έργο από ποια ακριβώς τρίτη χώρα θα προέρχεται το κατασκευαστικό, το δομικό υλικό. Και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ποιος μπορεί για εμάς. Ως αναθέτουσα αρχή, ισχύει μία σειρά νομικών ασαφιών στον τομέα αυτών και το ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι ε, εάν ένας υποψήφιος μπορεί να ζητήσει ε, νομική προστασία από ε, αυτόν τον κανονισμό και στην περίπτωση αυτή αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει σε, μεγάλη, σε πολύ χρονοβόρες διαδικασίες εξακρίβωσης. Επίσης, διαπιστώνεται πρόβλημα με τις υπερβολικά χαμηλές προσφορές και στην περίπτωση που εμείς τις επιτρέψουμε πρέπει να ενημερώσουμε τον υποβάλλοντα αυτήν την πολύ χαμηλή προσφορά και να τον ενημερώσουμε για την διαδικασία που θα επακολουθήσει. Για την διαδικασία δηλαδή εξακρίβωσης και για όλο το τυπικό που θα ακολουθηθεί. Και, το, και ο κίνδυνος ο κίνδυνος που υπάρχει σε αυτό είναι να ακυρωθεί η σύμβαση από τις μεγάλες παρατάσεις. Τέλος, να σας πω ότι για εμάς ο κανονισμός αυτός έχει κίνητρα εμπορικά και πολιτικά, τα οποία δεν εξυπηρετούν τον σκοπό της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων όχι μόνο δημιουργείται μεγάλη γραφειοκρατία, δημιουργείται επίσης και μεγάλη νομική ασάφεια στην ε, εκτέλεση των ε, δημοσίων συμβάσεων. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, παρακαλώ να, σας ε, να σκεφτείτε όλ... τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε με τον κανονισμό αυτό, ακόμα και εκείνους που αφορούν τις ε, επιμέρους διατάξεις σας λέω ότι αυτό δεν γίνεται να εφαρμοστεί στην πράξη, ιδιαίτερα από την πλευρά του τελωνιακού δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος ε, ομιλητής είναι ο κύριος Αλέν Μπερζέρ, πρώτος αντιπρόεδρος της ε, Alstom. Και είναι στο γραφείο των Βρυξελών. Κύριε Άσρομ. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω στα γαλλικά. Παρ' όλα αυτά έχω, για να απλοποιήσω τη ζωή όλων, υποβάλει τα τις διαφάνειές μου στα αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Αυτό είναι καθοριστικό για μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αμοιβαιότητα, αυτό το εργαλείο που επιτρέπει την αμοιβαιότητα να αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να ψηφίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα σας εξηγήσω και γιατί. Πρώτον, αν μπορούσαν να λειτουργήσουν και οι διαφάνειες, όπως έλεγε ο κύριος Βουίλκοκ, μιλάμε για αγορές που και στη μεταφορά και στην ενέργεια και στη μεταφορά ενέργειας πρόκειται για δημόσιες αγορές. Εδώ η στρατηγική μας είναι να παρουσιάζουμε, αν θέλετε, ολοκληρωμένα συστήματα και να υποβαλόμαστε κάθε φορά στις οδηγίες και στις συμφωνίες για τις δημόσιες προμήθειες και συμφωνώ απολύτως με τον τελευταίο ομιλητή, ο οποίος παρουσίασε το περίπλοκο του θέματος, το πόσο περίπλοκο είναι να μπορέσει κανείς να λειτουργήσει με τέτοιες διαδικασίες. Σήμερα Μιλούμε για μεγάλες αναδυόμενες χώρες, αναδυόμενες οικονομίες. 60% των παραγγελιών μας προέρχονται από αυτές τις χώρες και πρέπει να σας πω ότι το σκηνικό αλλάζει ραγδαία. Πριν από δύο χρόνια η κατάσταση ήταν διαφορετική. Είναι λοιπόν για μας περίπλοκο να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις νέες αγορές, ενώ οι παραδοσιακές μας αγορές δεν γνωρίζουν την ίδια ανάπτυξη. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε με αυτές τις χώρες, αυτές τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, με τις οποίες δεν έχουμε ούτε διμερείς ούτε πολυμερείς συμφωνίες και τα περισσότερα από αυτά που επιτυγχάνουμε σε αυτές τις χώρες μας οδηγούν σε περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. 56% των εργαζόμενων της επιχείρησής μας βρίσκεται ακόμα στην Ευρώπη. Εξάγουμε λοιπόν από την Ευρώπη σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, από τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία και με την Ελβετία. Το 90% των δραστηριοτήτων μας που προέρχονται από την Ελβετία εξάγονται. Είναι ένα πραγματικό θαύμα. Όλες οι προσβάσεις λοιπόν που μπορούμε να πετύχουμε σε όλες αυτές τις εξωτερικές αγορές μας οδηγούν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής μας θέσης σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε ότι σήμερα γνωρίζουμε νέους ανταγωνιστές οι οποίοι προέρχονται από αυτές τις αναδιόμενες οικονομίες. Τους συγχαίρω. Πρόκειται για άτομα καινούργια, για επιχειρήσεις καινούργιες όπως η CNR, κινέζικες επιχειρήσεις ή την Ding Dong Fan. Πρόκειται για εταιρείε, για ονόματα που θα πρέπει να τα συνηθίσουμε, να τα γνωρίσουμε. Πρόκειται για αξιοσέβαστους ανταγωνιστές, οι οποίοι πλέον δεν χρειάζονται απολύτως καμία προστασία στις τοπικές τους αγορές. Κοιτάξτε την ανάπτυξη αυτών των κινέζικων επιχειρήσεων και βλέπετε τα δύο τελευταία χρόνια η κινέζικη ανάπτυξη είναι υπερδιπλάσια της δικιάς μας 7-9% ε, και δεν έχει καμία σύγκριση με την Siemens, με την Bombardier ή άλλες παραδοσιακές ε, επιχειρήσεις του κλάδου. Οι εταιρείες από την Κίνα είναι νέοι πρωταγωνιστές στις αγορές μας και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε σαν ε, εισάξιες ε, επιχειρήσεις και εγώ προσωπικά τους συγχαίρω. Τώρα, όσον αφορά παραδείγματο χάνει την Ιαπωνία, η οποία από το 1994 έχει υπογράψει την ε, συμφωνία Και βλέπουμε ότι πριν από 10 χρόνια όταν υπεγράφει η πρώτη συμφωνία, η πρόσβασή μας στην αγορά της Ιαπωνίας είναι 0,2%. Σήμερα παραμένει στο 0,2%. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Οι ανταγωνιστές μας όμως, οι Ιάπωνες, είναι παρόντες στις δικές μας αγορές. Έχουν ήδη πολύ σημαντικές επιτυχίες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Δεν είναι φυσικό όμως να μην υπάρχει αμοιβαιότητα και να μπορούμε και εμείς να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες, σε διαγωνισμούς στην Ιαπωνία. Και αυτό δεν γίνεται επειδή δεν είμαστε παρόντες. Εμείς, η επιχείρησή μου, ο Όμιλος Άλστομ είναι παρόν στην Ιαπωνία εδώ και έναν αιώνα. Και δεν είναι λογικό και φυσικό να μην έχουμε καμία δυνατότητα συνεργασίας όσον αφορά την Κίνα και τον Καναδά και ευχαριστώ την κυρία Σαρνές που είναι παρούσα εδώ γιατί η έκθεσή της για την Κίνα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Σε κάποιους από τους τομείς της δραστηριότητάς μας βλέπουμε η κατάσταση με τις χώρες αυτές να είναι διαφορετική. Είμαστε παρόντες, είμαστε τοπικοί, έχουμε τοπική παρουσία. Παρ' όλα αυτά όλες αυτές οι αγορές είναι για μας σχεδόν αδύνατον να τις χρησιμοποιήσουμε. Για την Κίνα, λοιπόν, για την Ιαπωνία έχουμε ελάχιστες δυνατότητες και βλέπουμε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δεν είναι βιώσιμη αν συνεχίσουμε χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Βελτιώνεται η κατάσταση. Εγώ άκουσα προηγουμένως τον ε, προηγούμενο μιλητή, ο οποίος είπε ότι αυτή η νέα συμφωνία θα βελτιώσει τα πράγματα πότε αύριο. Μα μονίμως αύριο περιμένουμε να αλλάξουν τα πράγματα. Στις Ηνωμένε Πολιτείε η νέα κυβέρνηση Ομπάμα πέρασε ένα νομοσχέδιο που προβλέπει ότι το τοπικό περιεχόμενο για να μπορέσει να συμμετάσχει κανείς σε μια προκήρυξη διαγωνισμού για τους σιδηροδρόμους χρειάζεται 100% τοπικό περιεχόμενο. Μα αυτό είναι ένδειξη ανοίγματο των αγορών από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν νομίζω. Όσον αφορά τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα, είναι σαφής η προτίμηση για τις τοπικές επιχειρήσεις. Το λεγόμενο τοπικό περιεχόμενο λαμβάνεται υπόψη και οδηγεί σε μια δυσκολότερη πρόσβαση για μας στις αγορές αυτές. Τι μπορούμε να κάνουμε. Είτε θα αποφασίσουμε να μην κάνουμε τίποτα και θα παραμείνουμε στο, στην παρούσα κατάσταση, η οποία για μας δεν είναι πλέον βιώσιμη, και στρέφομαι προς την Επιτροπή λέγοντας ότι πραγματικά αν αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Η Επιτροπή προτείνει κάτι που συμπεριλαμβάνει ένα εργαλείο που είναι το άρθρο 8, 9 και 10 ένα εργαλείο που βασίζεται ουσιαστικά στις διαπραγματεύσεις Συγχαίρω αυτούς που έχουν αναλάβει αυτές τις διαπραγματεύσεις και προσπαθούν να πείσουν τους ε, εταίρους μας να ανοίξουν τις αγορές. Όταν όμω πάω εγώ στην Ιαπωνία και λέω στους Ιάπωνες ανοίξτε τις αγορές σας, γιατί οι δικές μας αγορές είναι ανοιχτές για αυτά, πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαπραγματευτούμε, καθότι δεν έχουμε κανένα μέσο στη διάθεσή μας, κανένα εργαλείο. Αυτή λοιπόν η μακροχρόνια διαδικασία διαπραγμάτευσης μπορεί να προσφέρει ένα κίνητρο αρνητικό θα έλεγα, μια απειλή, κάτι που σίγουρα θα αποτελέσει έναν από τους λόγους που θα οδηγήσουν κάποια στιγμή στους εταίρους μας να ανοίξουν τις αγορές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα ένα εργαλείο που ίσως έχει πιο βραχυπρόθεσμες ε, επιπτώσεις και που βασίζεται στον χρόνο μιας διαδικασίας προκήρυξης διαγωνισμού. Πρόκειται για το άρθρο 6. Πριν δηλαδή ξεκινήσουν οι παραγγελίες, πριν εκτελεστούν οι συμβάσεις. Αυτό το άρθρο 6 παρουσιάζει λοιπόν για μας κάποια πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και αν ακολουθήσουμε τη διαδικασία άρθρου 8 προς να προμηθευτεί η μία δημόσια αρχή λέγοντάς τους ότι δεν θα έπρεπε να είχατε κερδίσει αυτό το διαγωνισμό κάτι το οποίο τους το λέμε πολύ αργά γιατί ήδη έχουν εκτελέσει το έργο. Ίσως λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις το άρθρο 6 είναι ένα αποτελεσματικό έργο για μας. Τελειώνοντας ήθελα να σας πω ότι το άνοιγμα των δημόσιων προμηθειών στους τομείς μας μεταφράζεται με περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη. Και το γεγονός ότι ο αστυνομικός στην Αγγλία κρατάει ένα γκλόμπ, αυτό δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιεί και συνέχεια. Χρειαζόμαστε όμως ε, και αυτά τα μέσα εκφοβισμού και απειλής. Ο κύριος Έντριτς μίλησε για τις ανησυχίες του, για τις ανησυχίες που έχουν οι αναθέτουσες αρχές. Θα πρέπει να δούμε τι δυνατότητες απειλών εκφοβισμού έχουμε. Θα πρέπει να ξαναδούμε τα κατώτατα όρια των 5 εκατομμύριων ευρώ και θα πρέπει να βρούμε και πιο απλοποιημένες διαδικασίες για τις αναθέτουσες συγγνώμη, αρχές. Η νομική ασφάλεια επίσης για την πρόσβαση στις αγορές είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και αυτό όχι γιατί μεταφράζεται με την βεβαιότητα ότι κάποιος θα μπορέσει να αναλάβει ένα έργο, αλλά για μία μικρομεσαία επιχείρηση, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όταν κάποιος έχει πρόσβαση σε μία αγορά, στην Κίνα, στη Βραζιλία, στην Ινδία, και αν ξαφνικά βρεθεί εκτός των αγορών, γιατί κάποιος πολιτικός αποφάσισε να δώσει πλεονέκτημα στις τοπικές επιχειρήσεις, στους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και σε αυτό αναφέρομαι όταν ομιλώ για νομική ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε τώρα να περάσουμε στη συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακούσατε αρκετές παρατηρήσεις, πώς απαντάτε. Ευχαριστώ καθηγητά Μορέιρα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή αλλά και τους εισηγητές, τους ομιλητές για τη συζήτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Αν μου επιτρέπετε θα περάσω κατευθείαν σε κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν και δεν θα εκφωνήσω μία ακόμα ομιλία γιατί νομίζω ότι είναι καλό να σχολιάσουμε ορισμένα από αυτά που ακούσουμε. Ίσως το καλύτερο είναι να ξεκινήσω με το σχόλιο του κυρίου Νίγλου ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ένα μοντέλο ε, για το να ανοίξουν παγκοσμίω ε, οι αγορές δημοσίων συμβάσεων. Ε, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι σωστό να κλείνουμε τις αγορές μας και να είμαστε προστατευτικοί. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τον υπόλοιπο κόσμο να υιοθετήσει και τα δικά μας πρότυπα, γιατί Κανείς ε, άλλος ε, στον κόσμο ε, δεν έχει τέτοια πρόσβαση στην αγορά. Εμείς προτείνουμε ανοιχτή πρόσβαση χωρίς καμία προϋπόθεση σε συμβάσεις μέχρι 5 εκατομμύρια. Δεν θέτουμε καμία ερώτηση, απλώς πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε ένα πολύ καλά ε, ζυγισμένο μέσο για να δείχνουμε και μια κίτρινη κάρτα όταν χρειάζεται, όταν εμείς δεν έχουμε ισότιμη πρόσβαση στις αγορές των άλλων. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ είπατε και εσείς, εξακολουθούμε να έχουμε πολλά μέσα τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια και ε, βλέπουμε να υπάρχει ανάληψη δράσης από Αμερικανούς, Κινέζους κτλ. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να παραμείνουμε εκεί που είμαστε σήμερα. Τώρα, συμφωνώ με τον αλλομιλητή ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλά τα δεδομένα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δεδομένα και συμφωνώ με το ότι ένα ποσοστό του ότι είναι δυνατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντικατοπτρίζεται τώρα γιατί ε, εμείς δεν ελέγχουμε τις ιατρικές εταιρείες όταν ελέγχονται από ξένες εταιρείες ενώ όλοι οι άλλοι το κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε να συζητούμε για πάρα πολύ ώρα για το θέμα των αριθμών, όμως η νομική κατάσταση είναι ξεκάθαρη ότι δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα να κάνει κάποιος ε, προσφορά σε κάποιες από τις, μεγαλύτερες, από τις αναδυόμενες χώρες, ούτε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, βέβαια, ε, αυτό δείχνει ότι η αγορά, για να αγοράσει κανείς ε, αυτοκίνητα, ε, παραδείγματο χάρη στην Κίνα ήταν ανοιχτή μέχρι πέρσι και από πέρσι είπαν ότι έπρεπε να αγοραστούν κινέζικα αυτοκίνητα στην Κίνα για τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Αυτή είναι λοιπόν μια τάση, δεν θα αναφέρω όλα τα παραδείγματα που βλέπουμε, δεν θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε προβολή του τι έχουμε σήμερα, γιατί σε πολλές χώρες η ικανότητα που δεν υπήρχε τώρα υπάρχει για τοπική παραγωγή. Και αυτό είναι καλό από μόνο του, γιατί αυτό μας επιτρέπει να πουλάμε μηχανήματα και εξοπλισμό όμως ε, δεν θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από μια τάση να κλείσουν τις αγορές δημοσίων συμβάσεων. Τώρα το κόστος ε, και τα ωφέλη συζητήθηκαν λεπτομερώς. Εμείς δεν θέλουμε μια κατάσταση όπου να γίνεται πιο δύσκολη η διαδικασία. Εμείς εδώ μιλάμε για μια πραγματική εξαίρεση σε αυτό το δόγμα, σε αυτό το πιστεύω, αλλά θα έρθω και πάλι στο κόστος. Είχαμε μια καλή παρουσίαση για τα πιθανά προβλήματα, θα επανέλθω. Όμως ε, η τιμή για τα πιθανά αντιποδοτικά μέτρα, νομίζω ότι υπήρξε κάποια υπερβολή στα όσα ακούσαμε. Καταρχήν ο λόγος είναι αρκετά σαφής. Ε, είχαμε ανοιχτές αγορές, ανοιχτή αγορά ενώ οι υπόλοιποι δεν έχουν κάτι τέτοιο και δεν ξέρω σε πόσους ε, από εσά ασκήθηκε πίεση από τα διάφορα λόμπι. Εμάς μας κατηγόρησαν για ένα μεγάλο προστατευτικό μέτρο εδώ, γιατί όλοι κατανόησαν ότι απλώς προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη συμφωνία για το ότι είναι δυνατό και για τα πιθανά δίμετρα, αν ε, δούμε πώς συμπεριφέρονται και οι άλλοι. Φυσικά πολλά εξαρτώνται από το πώς ε, θα δούμε τα ε, πράγματα και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό θέλουμε από την Κομισιόν. Αν δείτε τον κανονισμό και τον τρόπο που τον έχουμε διαρθρώσει, αν υπάρχει κοινοτική δράση, έχουμε ε, έρευνα Έχουμε πολύ χρόνο για τις διαπραγματεύσεις. Ε, θα οικοδομήσουμε όλες τις πιθανές γέφυρες, τις δυνατές γέφυρες με τις άλλες χώρες πριν να σκεφτούμε μια κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και πολιτικό κόστος. Αλλά ήθελα να σας υπενθυμίσω, όταν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά την κρίση προέβησαν σε κλείσιμο των αγορών, ε, όταν ε, οι Κινέζοι έκαναν το ίδιο, δεν ανησυχούσαν για τα αποδοτικά μέτρα, γιατί ξέρουν ότι σε αυτό το στάδιο εμεί δεν έχουμε μέτρα να κλείσουμε τι δικέ μα αγορέ, ούτε καν νομική βάση δεν έχουμε. Θα λειτουργήσει. Και πάλι αυτή είναι η ερώτηση που τέθηκε από τον κύριο Χούλκοκ. Υπάρχουν ε, κάποια αποδεικτικά στοιχεία ότι κινούμαστε θετικά. Δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά στι διαπραγματεύσει που έχουμε για τι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με χώρε όπω ο Καναδά, όπω η Ινδία, βλέπουμε να υπάρχει κάπως μεγαλύτερη βούληση να σταθμίσουν τις πιθανές συνέπειες να μην διαπραγματευτούν κάτι καλό για τις δημόσιες συμβάσεις. Πιστεύω ότι έχουμε μία πρόταση επιτάπητος. Κατά την άποψή μου σίγουρα βοηθάει γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον υπάρχει κάτι σοβαρό που λαμβάνει η χώρα. Φυσικά δεν του έχουμε πείσει όλους και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, αλλά νομίζω ότι θα λειτουργήσει αν χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό με σοφροσύνη και με έναν τρόπο που θα βελτιώσει την κατάσταση σε πολλά μέρη του κόσμου. Αν έχω λίγο χρόνο, να επανέλθω και στο ότι αν ο νέος εξοπλισμός για τις διπλή αν είναι πάνω από 5 εκατομμύρια, μου φαίνεται κάπως ακριβώς, δεν ξέρω, αλλά αν είναι πάνω από, πάνω από αυτό το κατόφλι, αν θα είναι πιο δύσκολη η κατάσταση. Η απάντηση είναι, εξαρτάται από το πόσο συχνά οι τοπικές οντότητες θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. Εμείς εκτιμούμε όχι πολύ συχνά. Επειδή ε, γίνεται μια αναταραχή σε τοπικό επίπεδο, δεν θέλει να το χρησιμοποιήσει κανεί, εκτό και αν έχει πολύ καλούς λόγου. Αυτό σημαίνει ότι ε, στη δική τη περιφέρεια θα υπάρχει μια εταιρεία που παράγει το ίδιο προϊόν και θα είναι άδικο να μην προστρέξει κανεί αυτή την εταιρεία. Όμω αυτή δεν θα είναι πάρα πολύ συχνά. Ε, δεν θα είναι μια περίπτωση που θα τη συναντάμε πολύ συχνά. δεν ε, θα πρέπει να δουν ε, τον τελειωνιακό κώδικα, απλά θα πρέπει να ζητούν μία δήλωση από τον υποβάλλοντα προσφορά. Νομίζω ότι δεν θα είναι πολύ δύσκολο να λάβει κάποιο αυτή τη ε, δήλωση και οι εταιρείε που κάνουν προσφορές για συμβάσεις για πάνω από 5 εκατομμύρια θα είναι πολύ πιο εύκολο να δουν από πού προέρχονται τα προϊόντα. Νομίζω ότι αν μιλάμε για τέτοιες εταιρείες, ε, τότε σχετικά εύκολα αυτές, ε, επειδή θα έχουν μεγάλο τζίρο, θα μπορούν να πούν ναι ή όχι. Συχνά είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Χρησιμοποιούμε το κατόφλι ε, στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων. Δεν είναι το φίβραμε τώρα. είναι οι γενικοί κανόνες ε, που ισχύουν ε, για να δούμε τι ισχύει για τις προσφορές. Συμφωνώ ότι θα καθυστερήσουμε κάπως, μπορεί να χρειαστούμε δύο μήνες ή και τέσσερις μήνες. Ίσως αυτό είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε συνολικά Αλλά αν έχουμε μία-δύο περιπτώσεις ε, στην Ευρώπη, νομίζω ότι δεν είναι πολύ ψηλό το τίμημα. Αν έχουμε μία-δύο περιπτώσεις ετησίως, θα το αντιμετωπίσουμε. Και στο κόστος όφελος, το κάνουμε αυτό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να πούμε, και αυτό προέκυψε και από τις παρουσιάσεις, κανείς δεν αμφισβήτησε τους αριθμούς του μελέτη αντικτύπου για το θετικό αντίκτυπο, που θα υπάρξει σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτές οι αγορές ε, μεγεθύνονται και επομένως ο δικό μας εξοπλισμός ε, αυτό παράγονται θα είναι σε ζήτηση. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό. Δημιουργούμε τις ευκαιρίες και πρέπει να βασιστούμε στην δική μας ανταγωνιστικότητα. Δεν έχω πολλά να πω για την παρουσίαση της Alstom. Δεν το κάνουμε αυτό για μια συγκεκριμένη εταιρεία, για μεγάλες εταιρείες. Το κάνουμε για τους τομείς για τους οποίους η μελέτη που έδειξε ότι υπάρχει πραγματική αγορά όπου έχουμε πλεονέκτημα ανταγωνιστικό. Έχουμε τις τηλεπικοινωνίες, τα αεροπλάνα. Τι θα σημαίνει τώρα ε, για τις πωλήσει του Airbus ε, αν αφήσουμε τη Βραζιλία και την Κίνα να πάρουν την πρώτη καθεδρία. Θα σταματήσω εδώ. Αν μου επιτρέπετε, θέλει να πει και ο συνάδελφος δύο λόγια από την ΓΑΜΑ ΜΑΡΚΤ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, λέει ο Πρόεδρος, δύο-τρία λεπτά. Θέλω να κάνω τρία σχόλια. Καταρχήν, Για να απαντήσω, ίσως είπα ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι περισσότερο ανοιχτή από άλλε ξένες αγορές. Διαφωνώ κάθετα με αυτή τη δήλωση. Εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Γιατί η ευρωπαϊκή αγορά σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ε, ξένων προσφερόντων είναι 100% ανοιχτή σήμερα. Όλοι μπορούν ε, να συμμετέχουν ελεύθερα στις δημόσιες συμβάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κερδίζουν τόσο πολλέ συμβάσει. αλήθεια είναι αυτό, αλλά ο λόγο είναι ότι οι ευρωπαϊκές ε, εταιρείε είναι πιο ανταγωνιστικέ από τους ε, ξένους. Και επίσης, ε, συχνά οι αγορές συμβάσεων δεν είναι ανοιχτέ 100% ε, και οι δικές μας επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάνε να ανταγωνιστούν σε εκείνες τις αγορές. Έτσι λοιπόν αν ε, χάνουν κάποια συμβόλαια, κάποια συμβάσεις φαίνεται σαν να είναι κλειστή η αγορά μας. Αλλά αν το δείτε από την άλλη σκοπιά οι ξένοι επενδυτές 100% μπορεί να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές δημόσιες συμβάσεις. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι αν διαπραγματευτούμε διεθνώς σε πρόσβαση στις αγορές συμβάσεων μπορούμε ε, να αντιμετωπίσουμε τις χώρες ε, με τις οποίες έχουμε διαπραγματευτεί καλύτερα με, σε σχέση με αυτές με τις οποίες δεν έχουμε διαπραγματευτεί. Σήμερα, σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, σήμερα ε, οι χώρες με τις οποίες δεν έχουμε διαπραγματευτεί μπορούν ε, ελεύθερα να συμμετέχουν στις δικές μας διαδικασίες γιατί έχουμε ανοιχτέ αγορές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε στις διεθνείς διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Πολύ καλά το είπε ο κ. Ε, Νίγκλε ε, και πρέπει να προσθέσω στι διαπραγματεύσει για την GPA. Αυτέ είναι οι συνθήκε υπό τι οποίε πρέπει να εργαστούμε, γιατί δεν έχουμε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα. Αν είχαμε αυτό το μέσο, θα ήμασταν 10 φορέ καλύτεροι, έτσι ώστε να ε, σημειώσουμε τη διαφορά μεταξύ όσων συμφωνούν μαζί μας και πόσο και με αυτούς που δεν συμφωνούν. Τώρα, για όσα είπε ο κύριος Χάιριξ συμφωνώ και οι σημερινές ε, εταιρείε πρέπει να δραστηριοποιηθούν βάσει αυτού του καθεστώτος, όμως πρέπει να πω ότι όλες οι συμβάσεις κάτω των 5 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι ε, για όλους ε, και τους ξένους προσφέροντες και αυτό σημαίνει ότι φτάνουμε στο 97% των συμβάσεων. Επίσης, οι οντότες μπορούν να δεκτούν ξένους υποβάλλοντες προσφορές, είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν αν θέλουν να αποκλείσουν ε, τους αλλοδαπούς. Αν θέλουν να τους αποκλείσουν μπορούν να το κάνουν. Έτσι λοιπόν αυτό εξαρτάται από αυτούς όταν θα μπουν σε μία πολύπλοκη κατάσταση, γραφειοκρατική κατάσταση. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε αν ε, στο 47% των συμβάσεων μπορούμε ουσιαστικά να ξεφορτωθούμε το διοικητικό άχθος. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτο ακούσουμε τα μέλη της Επιτροπής. Ας ακούσουμε την άποψη του συναδέλφου μας στην Επιτροπή ΙΜΚΟ, την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών, διότι εκείνη αυτή τη στιγμή ασχολείται με την αναθεώρηση των ε, κανονισμών για τις δημόσιες συμβάσεις στην εσωτερική αγορά. Κύριε Άγγελ, έχετε το λόγο. Πείτε μας τι κάνετε στην ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς πολύ θα θέλαμε να είχαμε συμμετάσχει. Μας δώσετε μόνο 1,5 άρθρο, μόνο. Γι' αυτό και εμείς απλώς θα γνωμοδοτήσουμε. Τέλος τελικά το ίδιο ίσως θα είναι με αυτό που θα είχαμε κάνει από την αρχή. Δεν θα μιλήσω λοιπόν για το εργαλείο αυτό, καθε που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Το έκαναν οι προηγούμενοι ομιλητές και η Επιτροπή σας έχει ήδη επεξεργαστεί το θέμα αυτό στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται λοιπόν εδώ να επαναλάβω πράγματα τα οποία τα γνωρίζετε. Καταρχήν θα ήθελα όμως να πω, για να σας δείξω ποια είναι η προσέγγιση της δικής μας Επιτροπής για το θέμα της αμοιβαιότητας. Αν κοιτάξει κανείς τους αριθμούς σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά την πρόσβαση των εθνικών αγορών σε σχέση με ξένους ε, φορείς, αλλοδαπούς που θέλουν να προσχωρήσουν, είναι 0,08% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αναπτυχθεί εκτός των συνόρων μας 0,08% και αυτό δεν είναι τίποτα. Οι λόγοι είναι γνωστοί και ο κύριος λόγος, ο κύριος λόγος είναι ότι εμείς ανοίξαμε τις αγορές μας και οι άλλοι δεν άνοιξαν τις αγορές τους. Και το ερώτημα είναι αυτό το εργαλείο αμοιβαιότητας, οι ρήτρε αμοιβαιότητας ή με ποιον άλλο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Η απάντησή μου είναι ότι δεν θα πετύχουμε κάτι τέτοιο με αυτόν τον τρόπο. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δείξουμε ότι δεν θέλουμε να παραμείνουμε στην παρούσα κατάσταση και να συνεχίσουμε να δεχόμαστε τα πράγματα όσοι έχουν. Γι' αυτό και όσον αφορά τις δύο προτάσεις οδηγίας για τις δημόσιες προμήθειες. Τις δύο οδηγίες επαναλαμβάνω και το δίκτυο αλλά και για τις εκχωρήσεις. Εμείς υιοθετήσαμε μια θέση που θα μας επέτρεπε από την αρχή η θέση σε ισχύ αυτής της οδηγίας να δραστηριοποιηθούμε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν συνεχίσουν να μας αρνούνται κάθε πρόσβαση στις δημόσιες προμήθειές τους. Και την ίδια ώρα οι ίδιοι χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουμε, δυνατότητες οι οποίες θα είναι λιγότερο δεσμευτικές από αυτές που μέχρι τώρα ε, ισχύουν τι πρέπει να κάνουμε και πώς έχει η κατάσταση. Η κατάσταση σήμερα, όσον αφορά την οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες στα δίκτυα, ζητά την αμοιβαιότητα, ενώ η γενική οδηγία δεν απαιτεί αμοιβαιότητα. Είπαμε λοιπόν, για να υπάρχει συνοχή, ότι θα χρησιμοποιήσουμε ακριβώς την ίδια διατύπωση με αυτή που υπάρχει στην οδηγία για τα δίκτυα και να την ενσωματώσουμε αυτήν την διατύπωση, αυτή την σύνταξη και στη γενική οδηγία. Να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η ίδια ακριβώς διατύπωση και στις δύο οδηγίες έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε μία κοινή αντίδραση όταν υπάρχει στρέβλωση ανταγωνισμού. Για την οδηγία που αφορά τα δίκτυα το Συμβούλιο συμφώνησε, όχι όμως και για την άλλη οδηγία. Θα δούμε λοιπόν πού τελικά θα καταλήξουμε σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης μεταξύ των δύο ε, νομοθετικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι σε δύο οδηγίες, οι οποίες ακόμα δεν έχουν μεταφερθεί και οι οποίες θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια το νωρίτερο το Μάιο του 2013. Θεωρητικά λοιπόν αυτές οι δύο οδηγίες μετά από δύο χρόνια, δηλαδή το Μάιο του 2015, θα θεσπίσουν και θα θέσουν σε ισχύ κάποιες διατάξεις αμοιβαιότητας έτσι ώστε να μπορούμε να προσφύγουμε κατά κάποιου ο οποίος δεν ε, ακολουθεί αυτήν την αμοιβαιότητα και θέλουμε να του περιορίσουμε την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά. Εσείς εδώ και μήνες ασχολείστε με το θέμα αυτό και επεξεργάζεστε το θέμα αυτό. Εμείς γνωμοδοτήσαμε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ και οι διατάξεις αυτές θα αντικαταστήσουν έτσι και αλλιώς επειδή ακριβώς πρόκειται για κανονισμό, θα αντικαταστήσουν τις οδηγίες που υπάρχουν και ε, θα τεθούν σε ισχύ. Εάν λοιπόν αυτές οι διατάξεις για την αμοιβαιότητα είναι καλύτερες από αυτές που υπάρχουν στην οδηγία για τις δημόσιες συμβάσεις, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε επισπεύσει λίγο την διαδικασία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Αν αυτός ο κανονισμός δεν προχωρήσει καθόλου για κάποιο λόγο, σε αυτή την περίπτωση, επειδή θα ενσωματώσουμε στην οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες αυτές τις δυνατότητες προσφυγής που δεν υπάρχουν σήμερα, κάτι παρόλα αυτά θα έχουμε πετύχει καλύτερο. Και αν ο κανονισμός καθυστερήσει, μεταξύ, και αν η οδηγία μεταφερθεί, η οδηγία για τις δημόσιες προμήθειες, σε αυτή την περίπτωση κάτι θα έχουμε στο μεσοδιάστημα. Τι λέμε λοιπόν εμείς. Και αυτό είναι άσχετο με αυτά που κάνετε εσείς εδώ. Από τη στιγμή που η δική σας επιτροπής και το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια υιοθετήσει αυτό το εργαλείο, αυτές οι διατάξεις θα αντικαταστήσουν όλες τις υπόλοιπες. Εάν αυτό δεν γίνει, ενδεχομένως, και θα δούμε πώς θα πάνε και οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, κάποιες παρόμοιες διατάξεις, όχι ταυτόσιμες, να ε, υπάρξουν και να ενστοματωθούν σε κάποιες τομεακές σε κάποια κείμενα που αφορούν τους επιμέρους τομείς. Καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε μια καλύτερη διαπραγμάτευση, χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική μας θέση. Δεν θέλουμε να είμαστε βίαιοι σε καμία περίπτωση, αλλά συμβολικά πρέπει να εκφράσουμε την πολιτική μας βούληση. Γι' αυτό και θελήσαμε να βάλουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και αυτό ε, είναι το μόνο που θέλαμε να κάνουμε. Πρόεδρος. Ας ακούσουμε τώρα την ε, άποψη της Επιτροπής ΔΕΒΕ, κυρία Σαρτζεντίνη. The, um, public procurement. Οι δημόσιες συμβάσεις χρησιμοποιούνται για την εσωτερική ανάπτυξη των ε, κρατών, για τοπική ή εθνική. Και γι' αυτό λόγο αυτό δεν επετεύχθη καμία ε, κανονική συμφωνία ε, στην ΕΓΚΑΤΣ για τις δημόσιες συμβάσεις και δεν είναι οι χώρες αυτές ε, μέλη κάποιων συγκεκριμένων κανόνων. Υπάρχουν ε, πολυμερείς κανόνες. Κατανοώ ότι εσείς επιθυμείτε να έχετε έναν κανονισμό ο οποίος θα στοχεύει προς την Κίνα ή προς την Βραζιλία και με τον κανονισμό αυτό οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στην αγορά δημοσίων συμβάσεων εκεί στην Κίνα, στη Βραζιλία και σε άλλες αντίστοιχες χώρες. Όμως, ο ορισμός που χρησιμοποιείται σε αυτήν την πρόταση είναι οι χώρες εκτός από τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Η Κίνα Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΩΣΑ για, ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης είναι ακόμα μια αναπτυσσόμενη χώρα, το οποίο σημαίνει ότι αν ακολουθήσουμε τον ορισμό αυτό, δεν στοχεύεται μόνο στην Κίνα ή στην Βραζιλία, αλλά την Ουατεμάλα, το Βιετνάμ, το Φίτζι, την ακτή Ελεφαντοστού και την, την της Γάζας, για παράδειγμα, ακόμα, και το Καμερούν, μια χώρα με την οποία έχετε αυτή τη στιγμή ε, σχέσεις εμπορικές, οι οποίες, ε, η οποία τώρα πρόκειται να υπογράψει και μία ενδιάμεση συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν ως ε, εκπρόσωπος της Επιτροπής ΕΝΤΕΒΕ σας λέω ας μην το ψηφίσουμε ακόμα. Ας εξετάσουμε τις δυνατότητες δημοσίων συμβάσεων σε μια χώρα όπως οι προαναφερθήσεις. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς στην Επιτροπή ΙΝΤΑ είναι πώς εσείς επιθυμείτε να ορίσετε ε, την αμοιβαιότητα στον δημόσιο συμβάσεις, στον κανονισμό αυτό, χωρίς να βλάψετε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχει ένας ολόκληρος κατάλογος τέτοιων χωρών που έχει συντάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και ένας ακόμα μεγαλύτερος που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν. Το ερώτημά μου είναι πού στοχεύουμε. Στοχεύουμε στο να ανοίξουμε τις άλλες ε, αγορές ή το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία να κλείσουμε τη δική μας αγορά. Και από αναπτυξιακή άποψη δεν υπάρχουν πολλές χώρες που ε, συμμετέχουν στις δικές, στη δική μας αγορά συμβάσεων. Σχεδόν καμία, όπως είπε και ο συνάδελφος. Αλλά εάν υπήρχε θεωρητικά μια τέτοια ευκαιρία ε, για μια αναπτυσσόμενη χώρα ε, να αναλάβει δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ θα το χαιρετήσω. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, κλείνουμε τις αγορές μας με δικαιολογία, αυτό ή τις ανοίγουμε. Τέλος, ε, να σας πω ότι ως μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης κατά λίγο εκεί που άρχισε δηλαδή. Θέλουμε, ε, θέλουμε να έχουμε σχέσεις με μια χώρα σαν την Κίνα, αλλά ο κανονισμός αυτός στοχεύει και σε πολλά περισσότερα. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μέσο δημοσίων συμβάσεων για να τονώσουν την εθνική τους ή την τοπική τους οικονομία. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα από την Επιτροπή Απασχόλησης, ο κύριος Ντόιτς. Τρία λεπτά έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Στιάσαμε στα ακόλουθα σημεία και θα σας αναφέρω τα συμπεράσματά μου. Καταρχάς να τονίσω ότι η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών ε, Υποθέσεων δίνει μεγάλη σημασία σε μια κοινωνικά βιώσιμη διαδικασία δημοσίων συμβάσεων σε όλα τα στάδια, σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων. Δεύτερον, για μας είναι πάρα πολύ συναμπικό η νομοθεσία για την απασχόληση και τα πρότυπα για την απασχόληση και στα κρατημέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να, να πλαισιώνονται από κανονισμούς και για τις δημόσιες συμβάσεις. Τρίτον, να συμμεριστώ την άποψη του συναδέλφου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι εδώ μιλάμε για, μια, για στόχους ανταγωνιστικούς, για στρατηγικούς ανταγωνιστικούς στόχους, οι οποίοι ε, μας καθοδηγούν και πιστεύω πως ο σημαντικότερος από αυτούς τους στόχους είναι να τροποποιήσουμε και να αλλάξουμε τον κανονισμό για τις δημόσιες συμβάσεις έτσι ώστε να συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο απλή απάντηση σε αυτό είναι το να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει μόνο η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού, αλλά και, και η απαλήφη των ε, προτύπων και των κανονισμών που είναι βλαβεροί προς αυτό. Αυτό λοιπόν εμάς μας αναγκάζει να ξανασκεφτούμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιστεύω πως ε, θα πρέπει να δούμε ποια στοιχεία εργατικού δικαίου καθιστούν μειονέκτημα ε, μάλλον αποτελούν μειονέκτημα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να εισέλθουν αυτές τις αγορές των ε, τρίτων κρατών. Υπάρχει μια συμμετρία όσον αφορά τους ε, όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις αυτές. Μιλήσατε για αμοιβαιότητα αρκετά. Και όντως, η αμοιβαιότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι και ένα καλό μέσο για να επιτύχουμε το στόχο Uh, Μάλιστα, τώρα ανοίγουμε τη συζήτηση στην Επιτροπή, αρχίζοντας από τον εισηγητή κύριο Κασπάρη από το ΕΛΚ. Έχετε το λόγο. Ähm, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ομιλητές που πήραν το λόγο σε αυτή την ακρόαση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή τους. Ευχαριστώ πολύ και τους συναδέλφους που παρουσίασαν τη γνωμοδότηση των Επιτροπών. Καταρχήν να πω τρία πράγματα. Αυτό που είπε η Επιτροπή όσον αφορά τις 60.000 θέσεις εργασίας που είναι η επίπτωση αυτό κατά την άποψή μου, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ που έχω αυτή την άποψη. Δεν δικαιολογείται αυτός ο αριθμός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους αριθμούς με την ε, μελέτη αντικτύπου που έγινε. Εγώ θα ήθελα να μας εξηγήσει λοιπόν η Επιτροπή πώς, πού και με ποιο τρόπο έφτασε αυτό το αποτέλεσμα. Κύριε Μπουλοκ, άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε και αν κατάλαβα καλά αυτά που είπατε, είπατε ότι η εσωτερική αγορά θα έπρεπε να ολοκληρωθεί με καλύτερο τρόπο, να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή, αν θέλετε, και ότι οι ξένες επιχειρήσεις που βρίσκονται εδώ θα πρέπει να τους δοθούν καλύτερες προϋποθέσεις. Εγώ έχω πολλά παραδείγματα, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ που έχει τέτοιες ε, αν θέλετε, περιπτώσεις, όπως παραδείγματο χάρη το θέμα των γερμανικών σιδηροδρόμων και την χρησιμοποίηση του τούνελ κάτω από τη μάχη. άλλα παραδείγματα που αφορούν ε, την περιοχή μου που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με την ε, Γαλλία, κοντά στην Αλσατία δηλαδή και τη δυνατότητα συμμετοχής ε, επιχειρήσεων από την περιοχή μου στην διαδικασία διαγωνισμού, στην προκήρυξη διαγωνισμού στη Γαλλία. Πρόκειται για μια διακήρυξη που έγινε στα γαλλικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ το συγκριτικό πλεονέκτημα των γαλλόφωνων επιχειρήσεων ήταν προφανές. Τρίτο παράδειγμα, θα ήθελα να αναφερθώ στον συνάδελφο από την ΙΜΚΟ, ο οποίος αναφέρθηκε στην οδηγία για τις υπηρεσίες κοινή ωφελίας και εγώ θα ήθελα εδώ να μας αφήσει το θέμα αυτό, γιατί θεωρώ σαφέστατο ότι πρόκειται για θέμα δικής μας αρμοδιότητας. Τώρα, όσον αφορά τους ομιλητές, έχω κάποιες ερωτήσεις. Κατάλαβα ότι υπάρχουν εδώ διαφορετικές απόψεις και αξιολογήσεις όσον αφορά το κατά πόσο είναι ή δεν είναι αρκετά ανοιχτές οι αγορές μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικές αξιολογήσεις φτάνουν σε διαφορετικά αποτελέσματα. Κάποιοι λένε ότι το 60% των αγορών είναι ανοιχτό, άλλοι λένε 80% ή και παραπάνω. Θα ήθελα πραγματικά να κατανοήσω πώς φτάνουμε σε αυτά τα αποτελέσματα, ενώ βλέπουμε ότι η κατάσταση σε άλλες αγορές του κόσμου είναι τελείως διαφορετικά και στην πράξη στην πράξη υπάρχει η πραγματική πρόσβαση σε αυτές τις αγορές. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέμε ότι οι αγορές μας είναι ανοιχτές κατά 80%. Την ίδια ώρα όμως βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν ε, προσφορές από μέρους ξένων επιχειρήσεων. Η κινέζικη αγορά λέμε ότι είναι κλειστή, ενώ την ίδια ώρα γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν πολλές ε, επιχειρήσεις ε, που δεν είναι κινέζικες μπόρεσαν να εγκατασταθούν και να έχουν πολύ καλές ευκαιρίες και δυνατότητες. Αυτό λοιπόν αναφέρω όταν λέω στην πράξη ανοιχτές, πραγματικά ανοιχτές. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 58 και 59, ακούσαμε πολλά για αυτά τα δύο άρθρα. Γιατί όμως ποτέ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα αυτά τα δύο άρθρα. Η πρόταση της Επιτροπής ουσιαστικά κατά την άποψή μου μοιάζει πάρα πολύ η σημερινή πρόταση της Επιτροπής με αυτά τα δύο άρθρα, 58 και 59. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν γιατί εδώ και 10 χρόνια ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι δυνατότητες, μήπως είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν χρησιμοποιούνται ποτέ αυτά τα δύο άρθρα. Τρίτο ερώτημα. Η Επιτροπή αναφέρεται σε κάποιες εκτιμήσεις όσον αφορά το άρθρο 6, λέγοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 35 ή και παραπάνω φορές το χρόνο. Μπορείτε να μου πείτε πώς φτάσατε σε αυτήν την εκτίμηση. Δεν καταλαβαίνω. Θα με ενδιαφέρε πολύ να ξέρω πώς στηρίζετε αυτούς τους αριθμούς, αυτά τα στοιχεία, αυτές τις εκτιμήσεις. Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις που θέλω να κάνω καταρχήν. Και επίσης ο τρίτος ομιλητής αναφέρθηκε στο θέμα του γραφειοκρατικού βάρους, αναφερόμενος σε κάποιες συγκεκριμένες εκτιμήσεις, σε αριθμούς. Μήπως ε, μπορείτε να μου εκτιμήσετε πολύ συγκεκριμένα από πού φτάνουν αυτοί οι αριθμοί εθνικές ε, ρυθμίσεις ή εθνικές ε, νομοθεσίες που επιτρέπουν ή δεν επιτρέπουν την πρόσβαση στις αγορές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε ότι υπάρχει πραγματική συμβατότητα μεταξύ αυτών των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και κανονισμών και της ισχύουσας μέχρι τώρα ε, νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω τις ερωτήσεις μου η οδηγία της υπηρεσία κοινή ωφέλεια, το αρθρο 5859, το άρθρο 6, γιατί και πώς φτάνουμε στην εκτίμηση ότι μπορεί να χρησιμοποιεί 35-36 φορές το χρόνο και επίσης το θέμα του κόστους της γραφειοκρατίας ε, στον τελευταίο μιλητή. Σας ευχαριστώ πολύ. Well, uh, I hope... Πρόεδρος. Ελπίζω να σημείωσαν οι ομιλητές και οι κομισιόν τις ερωτήσεις ε, του εισηγητή. Ας ακούσουμε τους σκιώδεις. Ε, πρέπει να περιορίσω το χρόνο από εδώ και πέρα. από την ομάδα των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Τζιάν Λούκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές γιατί εμβάθυναν ιδιαίτερα στα θέματα αυτά αν και δεν συμφωνώ με κάποιε από τις σκέψεις τους. Εγώ παραμένω πεπισμένος ακόμη και μετά από αυτές τις ομιλίες για το πόσο σημαντική είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία όπως αυτή. Η πρώτη παρατήρησή μου έχει να κάνει με το εξή, ότι στο επίκεντρο τη προσοχή μα πρέπει να βρίσκεται η ευρωπαϊκή οικονομία και η ανταγωνιστικότητά τη. Το πρόβλημα και δυσκολίε των μέσων, όπω ε, αυτών που σχετίζεται με το δικαιωτικό κόστος και το γραφειοκρατικό άχθος ε, και επί των οποίων πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έρχονται στη συνέχεια. Τώρα στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσει, όχι ο μηχανισμός δημοσια διοίκηση. Θα πρέπει με βάση λοιπόν αυτά να νομοθετήσουμε. Μια ερώτηση που θέλω να θέσω και που ανέκυψε, αλλά θέλω να εμβαθύνω. Υπάρχουν πραγματικές εναλλακτικέ σε σχέση με αυτή που θέτουμε τώρα εμεί επιτάπητος και σε σχέση με τις προστατευτικές πρωτοβουλίες των υπολείπων. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι ένα υποκείμενο ε, που ουσιαστικά δεν ε, συμμετέχει στην ε, πραγματικότητα. Εμείς όμως δεν προβαίνουμε σε προστατευτισμό. Ζητάμε από τους άλλους να ανοίξουν τις αγορές τους και διατηρούμε ανοιχτέ τις δικές μας ε, και θέλουμε να δούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις τρευλώσεις στις δικές μας αγορές. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχουν εναλλακτικέ, ποιες είναι. Και αναφέρθηκαν κάποιες ε, χρήσιμες βελτιστές πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα κρατή-μέλη και που θα ήταν καλό να τις δούμε και εμείς. Μήπως μπορείτε να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες γι' αυτό. Τρίτον, κύριε να καταλάβω τουλάχιστον ε, συμφωνείτε για τον αυτόματο αποκλεισμό και πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Μία τελευταία παρατήρηση σε σχέση με τον αντίκτυπο στην απασχόληση. Εγώ κατάλαβα 60.000, όχι 600.000, γιατί μεταξύ των δύο αυτών αριθμών υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Όμως αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη ακόμη και 60.000 θα ήταν πολλές θέσεις εργασίας για αυτό το φαύλο κύκλο που μειώνουμε. Και επίσης πρέπει να δούμε και το θέμα της αμοιβαιότητας. Θα σταματήσω εδώ, γιατί έγινε και από τις παρατηρήσεις ε, και από τον κύριο Κασπάρη και από τους συναδέλφους ε, της ΣΥΜΚΟ. Εγώ συμφωνώ με κάποιες παρατηρήσεις του κύριου Κασπάρη και σας ευχαριστώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ο κύριος Κάζακα από το Άλντε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους ομιλητές για τη συνεισφορά τους σε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ιδίως ε, τον εκπρόσωπο της Alstom και τον εκπρόσωπο από τη Γερμανία. Ως και από τους φιλελευθερούς θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό. Φυσικά οι δημόσιες συμβάσεις είναι ένας πολύπλοκος φάκελος ε, παρά την επιδημία της Κομισιόν ε, να σπρώξει προς την απελευθέρωση των αγορών αυτών να γνωρίζουμε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις αγορές παραμένει γενικά κλειστή στις ευρωπαϊκές εταιρείες ε, που κάτι που έχει αντίκτυπο ε, για τις ε, εταιρείες σε κάποιους ε, τομείς πολύ σημαντικούς όπως οι μεταφορές και ο τομέας της ενέργειας. Έτσι λοιπόν μέχρι τώρα δεν είχε την κατάλληλη ε, εκτεταμένη πολιτική στον τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζουμε λοιπόν το νομοθέτημα αυτό και ελπίζουμε ότι αυτό το μέσο θα μας επιτρέψει να έχουμε διαπραγματευτεί πολιτικές ε, δυνατότητες έτσι ώστε να ασκήσουμε πίεση τη στιγμή ε, αυτή είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές. Υποστηρίζω λοιπόν την ιδέα του να έχουμε ένα εργαλείο αμοιβαιότητας στην διαδικασία του άρθρου 8 8-11 που είναι η διαδικασία ανοίγματο των αγορών. Το άρθρο 6 αντίθετα θα μπορούσε να ζημιώσει σημαντικά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση του προστατευτισμού. Θέλω μια ερώτηση να απευθύνω στην Κομισιόν για την έλλειψη ουσιαστική αμοιβαιότητα που ήταν το καθαριστικό κριτήριο για την επιβολή περιοριστικών μέτρων κατά τρίτων χωρών. Πώ ε, θα ήταν δυνατόν να αξιολογήσουμε το βαθμό διαφάνεια ε, χωρών και τη νομοθεσία για τι δημοσίε συμβάσει με τα διεθνή πρότυπα και πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει το βαθμό των διακριτικών πρακτικών κατά των υπηρεσιών ή των αγαθών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να καθορίσει αυτή την έλλειψη ουσιαστικής αβεβαιότητα. Επίσης, αναγνωρίζω τον πιθανό κίνδυνο ανταποδοτικών μέτρων που σχετίζονται με το μέσο, αλλά πιστεύω ότι ένας ισορροπημένος κανονισμός που θα μπορεί να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τις σημερινές στρατηγικές για την εκβιομηχάνηση και να αυξήσει το διαπραγματευτικό πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν θα συνεργαστώ με τον εισηγητή και τους όλους συναδέλφους για να διασφαλίσω ότι αυτά θα υπάρχουν στο τελικό κείμενο του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζαντόπο, τους Πρεσίρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να περιβρεθώ στις παρουσιάσεις. Είχαμε μια συζήτηση με τον Επιτροπό Ντεγκίχτ. Από αυτά που ακούω και από αυτά που μου οδηγήθηκαν... Πώς είπε ο εκπρόσωπο της Αριστούμενου, ερωτήθηκε ε, για ένα ποσοστό δημοσίων συμβάσεων που σήμερα είναι κλειστές και κυρίως για τους σιριοδρόμους και 100% σε ορισμένες χώρες. Αναρωτιέμαι, σε ποιο βαθμό η Alstom ε, μπόρεσε ή δεν μπόρεσε να υποφεληθεί από δημόσιε συμβάσει στη Γαλλία και στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια τη ύπαρξή τη. Η Alstom ε, σήμερα θα ήταν η Alstom χωρί δημόσιε συμβάσει. Τι θέλω να πω δηλαδή, εγώ κατανοώ το θέμα των δημοσίων συμβάσεων ε, και η αναθεώρηση να γίνει ευκαιρία για περαιτέρω αμοιβαιότητα. Εδώ συμφωνώ, αλλά ε, σήμερα όταν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ε, δεν θέτουμε την ερώτηση αν οι δημόσιες συμβάσεις είναι επίσης ένα εργαλείο βιομηχανικής πολιτικής αναρωτιέμαι για τη βούλησή μας ως Ευρωπαίοι ε, για να υπάρχει εξέλιξη των βιομηχανικών μας ικανοτήτων. Ξέρουμε ότι οι δημόσιες συμβάσεις ιστορικά και είναι λογικό αυτό γιατί ένα μεγάλο μέρος σχετίζεται με τα χρήματα του φορολογουμένου ήταν ένα μέσο ανάπτυξης μιας σειράς τομέων όχι απαραίτητο να αναθεθεί μία σύμβαση στο γειτονά μου, στο φίλο μου, ε, στον κουνιάδο μου, αλλά υπήρχε πραγματικά βιομηχανική φιλοδοξία πίσω από αυτό και ε, η Γαλλία και κάποιες άλλες χώρες, ε, η Γαλλία για τα φωτοβολταϊκά βάζει ένα Made in Europe για να καταπολεμήσει την αθέμητο ανταγωνισμό από την Κίνα και μου φαίνεται είναι, είναι νόμιμο αυτό, είναι και αυτή η βιομηχανική ιστορία. Κάποια στιγμή, κάποιοι τομείς να έχουν ανάγκη να υποστηριχθούν. Ειδικά όταν ξεκινούν και ειδικά όταν μιλάμε και για τοπικό επίπεδο να δώσουμε προτεραιότητα σε μικρές και μεσές επιχειρήσει, σε πολύ μικρέ επιχειρήσει σε μεσές επιχειρήσει σε επιχειρήσεις κοινωνικής και λιλέγγυης οικονομία, παρά στι πολυεθνικέ. Και δεν φτάνουμε σε αυτή τη συζήτηση αν θα ήταν επίση ενδιαφέρον εν δυνάμει να έχουμε και το τοπικό, τη τοπική συνιστόσα ε, και να, τε, αναλάβουμε. Γιατί όλοι το κάνουν αυτό και η Γερμανία και η Γαλλία, όλες οι χώρες. Αλλά όταν δεν αποδεχόμαστε ότι πρόκειται πραγματική διάσταση της βιομηχανικής πολιτικής μας, θεωρώ ότι είναι κρίμα. Και με εκπλήσει που η Άρστον σήμερα Καταλαβαίνω ότι θέλει να πάει σε όλε τι αγορέ, αλλά χωρί δημόσια συμβάσεις η Alstom ε, μάλλον δεν θα υπήρχε σήμερα. Ε, um, Χέλμουτ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω και τους ε, ομιλητές για τις παρουσιάσεις τους Τώρα, όσον αφορά την ε, να ασχοληθούμε περισσότερο με το θέμα. Πιστεύω πως είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα και ε, πέρα από όλα αυτά που σημειώθηκαν, που υπόθηκαν να πω και κάποιες άλλες απόψεις που για μένα δεν έχουν αναφερθεί ακόμα. Ε, για μένα είναι ζήτημα δημοκρατίας καταρχάς. Μιλάμε για πολυμερείς σχέσεις, μιλάμε για διμερείς σχέσεις, για τις δημόσιες συμβάσεις, όμως αυτό συμπεριλαμβάνει και εκείνους που βρίσκονται στο τέλος, αυτούς που πλήττονται, τους καταναλωτές. Και πρέπει να δούμε πώς εκείνοι θα παραλάβουν και θα απολαύσουν αυτές τις υπηρεσίες τέλος πάντων που θα προέρχονται από μια ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Και αυτό είναι πολύ περίπλοκο, το ε, πολύ περίπλοκο θέμα, ε, διότι αυτή η οδηγία έχει και σχέση με την οδηγία για τις παραχωρήσεις. Και εδώ αφορά και την ε, ενιαία αγορά το θέμα και το διεθνές εμπόριο. Και προσωπικά να το επαναλάβω το θέμα της ε, δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα τώρα ε, για εκείνους που ασχολούνται με το σχέδιο της ε, οδηγίας αυτής, διότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία σε ορισμένα σημεία. Υπάρχει κίνδυνος σε τοπικό επίπεδο που πλήττει τους πολίτες άμεσα και Όσον αφορά αυτά που είπε ο συνάδελφος Χάινριχ, σας καλώ να τα πάρετε στα σοβαρά. Πώς θα αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου μια περιφέρεια, μια κοινότητα, μια χώρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανταπεξέλθει σε έναν παγκόσμιο ανταγωνισμό εάν τηρήσουμε την αρχή αυτή που περιγράφεται. Πώς θα οργανώσουμε λοιπόν αυτόν τον ε, διαγωνισμό. Η οδηγία έχει ως σκοπό να ρυθμίσει, να ελέγξει και να επηρεάσει ε, τον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Ακούσατε τι είπαν οι συνάδελφοι για τους συνδυροδρόμους, ακούσατε για την ενέργεια, για, την, ε, για το νερό. Και όλα αυτά, πιστεύω, δεν έχουν ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην σύσταση της, ε, της ε, οδηγίας αυτής. Όσον αφορά την ε, πολυμερή διάσταση και για την Κίνα, των δισεκατομμυρίων, του 1,5 σχεδόν δισεκατομμυρίου κατοίκων. Τι θα γίνει αν εκείνοι θέλουν να συμμετέχουν, ας πούμε, σε μία σύμβαση εδώ σε ευρωπαϊκό έδαφος με πολύ λιγότερους κατοίκους. Πρέπει να δούμε την αναλογία της ε, ανάθεσης ε, παραχωρήσεων, της ε, ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και να δούμε, να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει αμοιβαιότητα και να μην υπάρχει ανεξέλεκτος ε, περιορισμός. Τέλος, να, να πω ότι όπως είπε και η αντιπρόσωπος της Επιτροπής Απασχόλησης, το ζήτημα της ε, απασχόλησης είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό στην οδηγία. Πρέπει να ακολουθήσουμε τα προστάγματα της, ε, της ε, Παγκόσμιας Χάρτας και να υιοθετήσουμε το κείμενο αυτό. Αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμεληθεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Γιάννικ Ραντό. Τι μας λέει. Πρέπει να δούμε τις δημόσιες συμβάσεις σαν εργαλείο της πολιτικής που υιοθετούμε. Συμφωνώ, συμφωνώ να υιοθετήσουμε μια νομοθεσία που να δίνει κάποια εκτίματα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, στις τοπικές επιχειρήσεις. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι έχουμε μια ανοιχτή αγορά, ιδιαίτερα για τις δημόσιες προμήθειες σε ξένες επιχειρήσεις, στον οποίο τις αγορές οι δικές μας επιχειρήσεις δεν μπορούν να μπουν. προς το παρόν η δική μου αγορά είναι ανοιχτή. Εξ των πολιτικών, τις οποίες στηρίζουμε εδώ και χρόνια και οι οποίες τελικά, κατά την άποψή μου, δεν είναι πάρα πολύ καλές, καθότι αν δει κανεί την κατάσταση όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη, προφανώς αυτή η πολιτική δεν είναι πάρα πολύ καλή. Όσον αφορά τον διεθνή ανταγωνισμό, είτε θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχωριστούμε τις δημόσιες αυτές συμβάσεις, είτε να υιοθετήσουμε κάποιους άλλους κανόνες, είτε να υπάρχει ανταγωνισμός πραγματικός και χωρίς καμία στρέβλωση. Γιατί σήμερα αφήνουμε, παραδείγματος χάρη, προϊόντα να μπαίνουν στην αγορά μας, προϊόντα τα οποία παράγονται με τελείως διαφορετικές προϋποθέσεις και περιορισμούς από αυτά που επιβάλλουμε στα προϊόντα που παράγονται στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να δημιουργούνται πολύ μεγάλες γιγάντιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα δεν ε, εμποδίζουμε στην Ιαπωνία, στην Κίνα και σε άλλες περιοχές του κόσμου να δημιουργούνται τέτοιοι γιγάντιοι όμιλοι επιχειρήσεων. Η αμοιβαιότητα λοιπόν δεν πρόκειται να ρυθμίσει όλα τα προβλήματα, αλλά πώς μπορούμε εδώ να αναρωτηθούμε αν είναι καλό αυτή η αμοιβαιότητα για τις εμπορικές συναλλαγές. Η απάντηση είναι σαφέστατη. Ναι, η αμοιβαιότητα είναι καλή, παρόλο που δεν αρκεί για μια καλή βιομηχανική πολιτική. Πρόεδρος. Eine ganz kurze Bemerkung. Ich bin... Πολύ σύντομα. Εγώ είμαι στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και δεν έχω πίστη ακόμα αν είναι λογικό ή δεν είναι λογικό αυτό που πάμε να κάνουμε. Και θεωρώ ότι αυτή η ακρόαση θα μπορούσε να μας βοηθήσει, τελικά όμως εμένα δεν με βοήθησε. Και πιστεύω ότι το θέμα το εμπορικό της εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει να συζητηθεί με πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την εσωτερική αγορά. Παραδείγματος χάρη, οι κοινότητες θα πρέπει να μπορούν να συζητήσουν με τους πολίτες που ζουν σε αυτή την περιοχή, που ψηφίζουν εκεί για το τι θέλουν να κάνουν και κατόπιν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις και να προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κριτήρια περιβαλλοντολογικά και καινοτομία. Αλλά, κύριε Σόλτς, οι ρυθμίσεις, οι κανονισμοί είναι κάτι που το αποφασίζουν οι κοινότητες και όχι οι Βρυξέλλες. Και αυτό, αυτή η αποκεντρωμένη προσέγγιση θα πρέπει να παραμείνει. Δεν μπορεί να αποφασίσει οι Βρυξέλλες για τη διαδικασία. Αυτό αποφασίζεται επιτόπου και με δημοκρατικό τρόπο. Και σε αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε. Ευχαριστώ και θα δώσω το λόγο στους ομιλητές. Αν θέλετε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, στις επιφυλάξεις. Και η Επιτροπή όμως θα πάρει το λόγο, γιατί ακούσαμε κάποιους αριθμούς, κάποιες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν για τρία λεπτά έχει το λόγο η Επιτροπή και μπορείτε να απαντήσετε στις παρατηρήσεις που σας έγιναν. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Ναι, όντως έγιναν κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, πού βρήκαμε αυτούς τους αριθμούς για τις θέσεις απασχόλησης. Αυτό τον αριθμό, αν θέλετε, τον υπολογίσαμε εμείς, δεν υπάρχει κάποιος ιδανικός τρόπος. Κοιτάξαμε τις εξαγωγές και είδαμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των εξαγωγών και των θέσεων απασχόλησης. Δεν πρόκειται για ακριβείς αριθμούς, αλλά έχουμε κάποια εμπειρία και πρέπει να σας πω ότι η ψαλίδα που χρησιμοποιήσαμε είναι η πιο χαμηλή και βεβαίως μπορούμε να δικαιολογήσουμε αυτούς τους αριθμούς. Για το 58-59, τα άρθρα αυτά που ρωτήσατε γιατί δεν χρησιμοποιούνται, γιατί δεν είναι σαφές το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Καταλαβαίνετε ότι κανείς μέχρι τώρα δεν το χρησιμοποίησε, είναι επικίνδυνο λίγο το έδαφος και γι' αυτό και πιστεύουμε δεν χρησιμοποιείται. Ας πούμε ότι αρχικά δεν είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και σήμερα προτείνουμε κάτι το πολύ πιο συγκεκριμένο και κάτι που εμπεριέχει και μια ευρωπαϊκή συνιστόσα, κάτι που δεν έχει η άλλη οδηγία. Τώρα, η έλλειψη ουσιαστικής αμοιβαιότητας. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση, γιατί θα πρέπει να κοιτάξουμε την ομοθεσία των χωρών στις οποίες αναφερόμαστε, να δούμε πολύ συγκεκριμένα τι ισχύει στην κάθε χώρα, να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση και αν θέλουμε να πάρουμε μια νομικά δεσμευτική απόφαση θα πρέπει να γίνει μια έρευνα επιτόπου για να δούμε για ποιο λόγο η πραγματική κατάσταση είναι αυτή, έλλειψη αμοιβαιότητας. Γιατί όπως ξέρετε άλλα συμβαίνουν τα κείμενα στην νομοθεσία και άλλα είναι, άλλη είναι πολλές φορές η πραγματικότητα. 35, 55 περιπτώσεις είπατε για το άρθρο 6. Θα απαντήσει ο συνάδελφος. Ναι, επίσης όσον αφορά τα κράτη-μέλη που έχουν νομοθετήσει επί του θέματος αυτού, όσον αφορά δηλαδή τη συμμετοχή ή μη στην προκήρυξη ενός διαγωνισμού, τι ισχύει και όπως ξέρετε η εσωτερική αγορά έχει υλοποιηθεί και οι πραγματικότητες δεν είναι πάντα οι στα κράτη-μέλη. Και εδώ σαφώς και θα υπήρχαν πολλοί λόγοι να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη εναρμόνιση. Κύριε Κάσπαρη, είπατε επίσης πώς φτάσαμε σε αυτόν τον αριθμό 35 με 50 περιπτώσεις ε, κάθε χρόνο. Δεν θα μπω τώρα σε όλες τις λεπτομέρειες, να σας εξηγήσω όμως. Καταρχήν, μόνο 7% όλων αυτών των περιπτώσεων, μόνο το 7% πρόκειται να ε, αναφερθούν στο άρθρο 6. Αυτό είναι κάτι Γιατί, διότι καταρχήν σε πολλούς τομείς όπως τα φάρμακα, τους υπολογιστές, οι τοπικές εθνικές αρχές δεν πρόκειται να αποκλείσουν τους, ε, τις ξένες επιχειρήσεις εξορισμού και εκ των προτέρων από τους διαγωνισμούς. Και ξέρουμε ότι αυτός ο αποκλεισμός δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάση του άρθρου 6 για τις πιο πολλές περιπτώσεις και πολύ λίγες θα είναι οι επιχειρήσεις αυτές που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που τους δίνονται είτε επειδή η γραφειοκρατία είναι τεράστια είτε επειδή θα υπάρχουν άλλα εμπόδια. Γι' αυτό και είπαμε ότι μόνο το 15 με 20% των περιπτώσεων θα αποκλείονται πραγματικά ε, και θα αποκλείουν πραγματικά τις ξένες επιχειρήσεις και μόνο αυτές μπορούν να μπουν στο άρθρο 6. Ευχαριστώ πολύ για τις διευκρινήσεις σας. Τώρα έχει έρθει η ώρα για τους ομιλητές με την ίδια Σειρά, τρεις, τρία λεπτό καθένας. Κύριε Νίλη. Ευχαριστώ. Θα είμαι περιπετειώδη και θα προσπαθήσω να κάνω μια παρέμβαση στη γλώσσα του Μολιέρου. Είναι ελβετική γλώσσα, δεν είναι, λέει ο πρόεδρος, βεβαίως. Έχω την εντύπωση και είναι μεγάλη ικανοποίηση αυτή ότι σε αυτή τη συνέλευση συμφωνούμε τουλάχιστον για ένα σημείο. Ότι δεν είναι αρκετά ικανοποιητικά τα πράγματα έτσι όπως έχουν. Αλλά θα ήθελα να καθησυχάσω εδώ μια σειρά μερών. Κινούνται τα πράγματα. Και μάλιστα δεν κινούνται ήδη από αύριο. Αν μου επιτρέπετε, η αλλαγή είναι τώρα και στον ΠΟΕ χτες. Δηλαδή το ότι έχουμε αυτό το νέο μέσο στον ΠΟΕ πραγματικά αλλάζει πάρα πολύ το τοπίο των δημοσίων συμβάσεων σε διεθνέ επίπεδο και πράγματι θα διευκολύνει αυτό που θέλουμε όλοι να θα διευκολύνει την κατάσταση και θα, μεγαλ... θα βοηθήσει στο άνοιγμα οι αγορές που είναι ανοιχτές de facto ή de jure είναι κάπως πιο πολύπλοκες αν ε, δούμε το θέμα από καθαρά νομική σκοπιά. Τώρα, για το, αν, ε, τώρα αυτό συμβαίνει επειδή de jure είναι κλειστές οι αγορές και δεν μπορούμε να μπούμε de facto, όχι. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπαίνουν σε αγορές που de είναι Τώρα, ε, αυτό είναι ικανοποιητικό, πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, δεν νομίζω. Πρέπει να πάμε σε δεσμευτική νομοθεσία και αν είναι δυνατόν και σε επίπεδο που ε. Για να μας καλύπτει και το όργανο επίλυσης διαφορών. Μιλήσαμε πολύ για τις αναδυόμενες χώρες στο στάδιο αυτό, οι δημόσιες προμήθειες που καλύπτονται από τα 40 μέλη του ΠΟΕ φτάνουν στα 1.603 δολάρια ετησίως. Εκτιμούμε ότι μία αγορά ενός δισεκατομμυρίου ε, ετησίως θα μπορούσε να ανοίξει αν συμμετείχαν όλοι σε αυτή τη συμφωνία, αλλά γιατί δεν το έχουν κάνει. Ε, η απάντησή μου είναι η εξή. Γιατί δεν ήταν ικανοποιητική η συμφωνία του 1995 ήταν ε, μια συμφωνία one size fits all, που να ταιριάζει για όλους, αλλά δεν τους ικανοποιούσε όλους. Τώρα, πώς θα καταπολεμήσουμε τις τάσεις προστατευτισμού. Και πάλι εδώ το πολυμερές ε, βήμα, το πολυμερές φόρουμ με την GPA δίνει μια καλή απάντηση, όπως ε, είδαμε για το Buy American. Κατάλαβαν οι Αμερικανοί ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό πια το Buy American. Κατανοούν ότι είναι καλύτερο να λένε Buy GPA αν υπάρχει εδώ ένας αντίκτυπος για τη βιομηχανική ικανότητα, δυναμικότητα και για τη δημιουργία θεσμών εργασία. Θέλω να σα πω ότι μεγάλε δημόσιε συμβάσει συχνά υποδιαιρούνται σε μικρότερα μέρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και φυσικά αυτό ωφελεί και τι ε, αλλοδαπέ και τι εγχώριε επιχειρήσει και τι μικρέ και τι μεγάλε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Και σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική τάση προς περισσότερη διακυβέρνηση. Σας παρακαλώ, μπορείτε να με μακρηγορείτε, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα, σα παραμείνουμε εδώ και τύπο στο διάδρομο θα συνεχίσω. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ο καθηγητής Γουλκοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ερώτημα του κυρίου Κασπάρη για το αν είναι οι αγορέ ανοιχτέ. Αν δείτε τα νούμερα και τα ποσοστά διασυνοριακών ε, αγορών στην Ευρώπη θα δείτε ότι είναι περίπου στο 45% των συμβάσεων. Και αν συμπεριλαμβάνετε και τις ε, και την προμήθεια από όλου τομεί, ανεβαίνουμε ακόμα περισσότερο στα ποσοστά. Και τώρα το θέμα ναι, είναι πώ το μετράμε. Αν δούμε τα, στοιχεία παγκοσμίω, θα καταλήξουμε σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Τώρα, σε συγκεκριμένου τομεί, ε, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για σημαντικέ συμβάσει, για παράδειγμα, ένα σιδηροδρομικό έργο που κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ και θα έχει μεγάλες ε, επιπτώσεις και συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα, δεν υπάρχει κάποια απλή απάντηση πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε και τα στοιχεία παγκοσμίω και τα στοιχεία ανά συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, μας είπατε ότι δεν υπάρχουν συμβάσεις που να πηγαίνουν και σε τρίτους αναδόχους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα χρήματα των φορολογούμενων για να αναθέτετε δουλειές ε, εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτό βέβαια είναι όντω μια δυσκολία στην αγορά των συμβάσεων. Πιστεύω πως ε, στο μόνο στο οποίο θα αλλάξει είναι αν υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση και εάν οι εταιρείε ε, σταματήσουν να έχουν μια αποκλειστικά εθνική ταυτότητα. Αυτό συμβαίνει και στην ενιαία αγορά, ας πούμε. Όταν χρησιμοποιούνται οι δημόσιες συμβάσεις για εθνικές πολιτικές, εκεί καταλήγουμε. Ποιες εναλλακτικέ ε, λύσεις έχουμε τώρα από το GPA. Πιστεύω πως, ε, και για να το συνδέσω κιόλα και με το ζήτημα της ανάπτυξης, πιστεύω ότι το GPA μας, ε, μας δημιουργεί μία δίωδο για μία πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση και δεν θα είναι εύκολο βέβαια για τις ε, χώρες να υιοθετήσουν μια πιο διάφανη μέθοδο ανάθεσης ε, δημοσίων συμβάσεων αλλά και όσο για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κάνουν και αυτή τη στιγμή αποθαρρύνονται από το να το κάνουν διότι δεν το βλέπουν ως αμοιβαιότητα. Είναι ένας κίνδυνος αυτός διότι θα, ε, θα πρέπει αυτές ε, οι χώρες βέβαια να έχουν κανόνες και νόμους, όμως αυτό από τη δική τους πλευρά θα θεωρηθεί ως ε, μία απλή δικαιολογία για την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα. Ότι δηλαδή δεν στοχεύουμε έτσι, στις αναπτυσσόμενες χώρες, δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να τις υπονομεύσουμε και νομίζω όμως πως δεν έχω χρόνο να απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις, οπότε θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος, ο κύριος Χάινριχ. Ο κύριος Κασπάρη ε, μίλησε για την εκτίμηση του διοικητικού κόστους. Ε, ναι, κύριε Κασπάρη, φυσικά δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και εξειδικευμένες αναλύσεις στον τομέα αυτό που να δείχνουν ποια είναι η σχέση του κόστους και της ε, πολυπλοκότητας των ε, διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. Όμως, η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξή. Οι δημόσιες υπηρεσίες χρησιμοποιούν ορισμένους ειδικού οι οποίοι ασχολούνται μόνο με το δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων και ασχολούνται με πολύ περίπλοκες διαδικασίες. Επίσης προσλαμβάνουν ειδικά, ειδικούς νομικούς που ασχολούνται με αυτό. Και ε, από αυτό μπορώ να σας πω ότι το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό. Και με τα, με τα μέσα που θα δημιουργήσει αυτός ο κανονισμός δεν θα μειωθεί. Τώρα θα ήθελα να πάρω την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα επιχείρημα που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, οι επιπτώσεις του κανονισμού για τις ε, δημόσιες συμβάσεις. Ναι, να σας πω ότι δεν θα το φάμε και καυτό. Θα περιμένουμε λιγάκι, διότι είναι πολύ σπάνιο να εφαρμοστεί άμεσα ο κανονισμός. Πρέπει να περάσει κάποιος ε, χρόνος. Να σας πω, για παράδειγμα, τι γίνεται με τα κατασκευαστικά έργα και τα μέτρα. Εκεί μπορούμε πολύ εύκολα να ξεπεράσουμε αυτό το κόστος ε, των 5 δισεκατομμυρίων που είπατε. Πάρα πολύ εύκολα. Με μία ανακαίνιση, για παράδειγμα. Και σε αυτόν τον τομέα των ε, κατασκευαστικών έργων, να πω ότι εκεί παρατηρούμε κατακαιρματισμό των συμβάσεων. Και αυτές γίνονται με προκήρυξη πανευρωπαϊκή. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ο κανονισμός έχει να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτές τις ε, περιπτώσεις, έχει να αντιμετωπίσει έχει να, πρέπει να δημιουργήσει μέσα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτού του κατακαιρματισμού και δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Σας ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος Μπερζέ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Κάσπαρη που αναφέρεται στο αν είναι κλειστές ή ανοιχτές οι ευρωπαϊκές αγορές. Είναι προφανές στην Ευρώπη ότι οποιοδήποτε θέλει να κοιτάξει την αγορά των δημόσιων συμβάσεων αρκεί να αγοράσει την εφημερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Υπάρχουν τα πάντα. Τα πάντα με πάρα πολύ σε κάθαρο τρόπο και με μεγάλη διαφάνεια. Αν θέλει να κάνει το ίδιο με την ε, Ιαπωνέζικη αγορά, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία δημοσίευση. Δεν υπάρχει τίποτα. Και αυτό το λέω ότι δεν είναι θέμα του αν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε ή όχι ένα διαγωνισμό. Απλώς δεν υπάρχει σαν έννοια η δημοσίευση των δυνατοτήτων να συμμετάσχει κανείς. Άρα κανείς δεν έχει καν τη δυνατότητα να γνωρίζει ότι θα προκηρυχθεί ένας τέτοιος ε, διαγωνισμός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, δεν είναι θέμα του αν ναι ή όχι οι αγορές είναι ανοιχτές, όταν κανείς δεν γνωρίζει καν τις δυνατότητες που υπάρχουν. Βεβαίως τα πράγματα δεν είναι ιδανικά και στην Ευρώπη, αλλά σήμερα κάτι άλλο συζητούμε. Κύριε Σαντό, νομίζω ότι η κυρία Σαρνέ σας απάντησε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ θα δεχόμουν ότι η βιομηχανική η πολιτική της Ευρώπης θα μπορούσε να υποστηρίζεται και να εξυπηρετείται από αυτήν την ε, συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις. Όμως σήμερα για μεγάλες χώρες, δεν αναφέραμε στη Μπουρκινα Φάσο ή στο Μάλι, σε μεγάλες όμως αναδιόμενες οικονομίες, οι οποίες διαθέτουν σήμερα ομίλους ισχυρούς που δεν χρειάζεται να στηριχθούν και να ενισχυθούν, όπως εμείς δεν χρειάζεται να ενισχυθούμε στις δικές μας αγορές, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει αμοιβαιότητα, διότι εκείνες οι εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτες και χωρίς ανταγωνισμό στις δικές τους αγορές, εμείς στις δικές μας αγορές θα πρέπει να μοιραστούμε τις δυνατότητες με επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να μας ανταγωνιστούν στην δική μας χώρα και στις δικές μας αγορές. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για το ένα ή το άλλο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής θέλει να κάνει κάποια τελευταία σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, τους κοιόδες εισηγητές, τα άτομα που εκπροσώπησαν τις άλλες επιτροπές με τις γνωμοδοτήσεις τους. Θα επανέλθει το θέμα, φαντάζομαι, στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και εκεί θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλοι μας μάθαμε πολλά. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των ακροάσεων. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο. Να επιτρέψουμε να αποχωρήσουν οι καλεσμένοι μας. Please, uh, the Σας παρακαλώ, θέλετε να συζητήσετε εκτός της αίθουσας.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 This is a, an opinion. για μια γνωμοδότηση για την ε, Ήτρα. Συντάκτρια της γνωμοδότηση η Μαρία Δεσσαρνές. Έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θα της δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσει το ζήτημα. Euh, Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να με ακρηγορήσω. Πρόκειται για μια πρώτη τελεγή απόψεων. Επομένως, ε, θα ήθελα να ακούσω τι θα πολλοί συνάδελφοι και οι σκιώδες εισηγητής αλλά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της Επιτροπής για ένα θέμα που σχετίζεται άμεσα με το προηγούμενο θέμα καθώς πρόκειται για την εκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Η διαπίστωση που πρέπει να κάνουμε από κοινού, καταρχήν πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό, είναι να δούμε την κατάσταση κατά πρόσωπο, να δούμε ότι στην Ευρώπη έχουμε χάσει 10 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη βιομηχανία τα 10 τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα τα 3 τελευταία χρόνια. Είχαμε μείωση της παραγωγής κατά 10% και χάσαμε 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στη βιομηχανία. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να έχουμε κατά νου. Η Ευρώπη ουσιαστικά είναι σε διαδικασία αποβιομηχάνησης, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο βλέπουμε να υπάρχει πρόοδος της βιομηχανίας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μας ικανοποιεί. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να το δούμε αυτό ως μοιραίο, αλλά για να μην γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή βούληση για το ζήτημα της βιομηχανοποίησης, χρειαζόμαστε πολιτική βούληση στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε μια πολιτική εκβιομηχανηση της Ευρώπης, μια κοινή πολιτική. Χαίρομαι που είδα λοιπόν το κείμενο της Κομισιόν που μας ε, δίνει κάποιους καλούς προσανατολισμούς. Η Επιτροπή προτείνει να διερευνήσουμε νέους ε, τομείς για την εκβιομηχάνηση. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Πρόκειται για νέους τομείς ε, στον τομέα μιας εκβιομηχάνησης, βιώσιμης και καθαρής και το θεωρώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς επί των οποίων σήμερα βρίσκεται σε κατάσταση χμής η Ευρώπη, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροναυπηγενική, το διάστημα, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα χημικά. Πρόκειται για τομεί όπου δεν πρέπει να εγκαταλείψει η Ευρώπη την προκαθεδρία. Πρέπει να τη διατηρήσει πέρα από τους ε, τομείς προτεραιότητας που αναφέρει η Κομισιόν, εγώ βλέπω και άλλους τομείς προτεραιότητας που είναι μεγάλες υποδομές μεταφορών, ενέργειας, τηλεπικοινωνίας. Φυσικά τίθεται το θέμα επενδύσεων και χρηματοδότησης και θα φτάσω και εκεί σε δύο λεπτά. Επίσης έχουμε το θέμα του στρατηγικού τομέα της ενέργειας. Όταν ε, βλέπουμε τις τιμές της ενέργειας και την αύξησή τους, ε, θα πρέπει να πούμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια κοινή ενεργειακή πολιτική και είναι δυνατόν θα πρέπει να κάνουμε να πέσουν οι τιμές στην ενέργεια και να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική στο θέμα. Θα μπορούσα να αναφερθώ και στο θέμα της βιοπιστικής βιομηχανίας. Είναι μια πολιτική, ένα τομέα που πρέπει να ενισχύσει η Ευρώπη, γιατί πρέπει να ενισχύσει την ανεκνευσιμότητα, θα μπορούσα να μιλήσω και για την άμυνα. Όλοι αυτοί οι τομεί δεν αναφέρονται καθόλου στην ανακοίνωση τη Κομισιόν, αλλά για μένα είναι στρατηγική τομή για το μέλλον. Και θα ήθελα να σας ε, πω ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός. Πιστεύω ότι καταρχήν τίθεται το θέμα των απαραίτητων επενδύσεων, των πόρων, των μέσων. Αν παραδείγματο χάρη δούμε την ανάπτυξη των μεγάλων υποδομών στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, που χρειάζεται η βιομηχανία τις επόμενες δεκαετίες, φτάνουμε περίπου στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και βλέπουμε ότι στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υπάρχουν δυσκολίες ε, και ε, υπάρχει μείωση του προπολογισμού. Έτσι λοιπόν, ε, να ρωτιέμαι μήπως θα έπρεπε για ορισμένα βιομηχανικά project να χρησιμοποιήσουμε το παθηματικό. Και επίσης πρέπει να δούμε και το θέμα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σήμερα δεν ε, μπορούν να βρουν εύκολα χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε το πρόβλημα με τις τράπεζες, με την τραπεζική πίστοση και δυστυχώς ε, τα χρήματα που υπάρχουν από τις τράπεζες στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορούν να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ίσως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να είναι μια απάντηση, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες απαντήσεις στην Τραπεζική Ένωση. Και Φυσικά υπάρχει και το θέμα των πολιτικών έρευνα και καινοτομία. Αν η Ευρώπη ε, θέλει να διατηρήσει πρωταρχική θέση, την προκαθερία θα πρέπει να αποκτήσει ε, ουσιαστικά και ε, μια ενίσχυση των πολιτικών αυτών. Δεν έχουμε επαρκή προπολογισμό, επομένως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαθέσουμε πόρους από τον εθνικό, τους εθνικούς και να υπάρχει καλύτερος συντονισμός. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεχνίας ήταν ένα καλό νέο, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει εγγύηση της προστασίας των διανοητικών δικαιωμάτων των επιχειρήσεων. Επίσης, ε, πρέπει να σκεφτούμε ε, και τη δημιουργία ευρωπαϊκών γιγάντων σε ορισμένου τομεί. Δεν ξέρω αν σήμερα η πολιτική ανταγωνισμού θα επέτρεπε να δημιουργηθούν ε, νέοι γιγαντέ, αλλά νομίζω ότι για το Airbus, παραδείγματο χάρη, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να ξαναδημιουργηθεί, αλλά ε, λυπάμαι που δεν έγινε συγχώνευση μεταξύ ADS και BA και νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο. Χρειαζόμαστε Ευρωπαίους πρωτεθλητές, ε, γίγαντες, είναι αυτό απόλυτα απαραίτητο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Και συνεχίζω με τον καταλογό μου, χρειαζόμαστε να εργαστούμε για την σήμανση προέλευσης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα είδατε το σκάνδαλο που ζήσαμε πρόσφατα στο γεωπιστικό τομέα και επίσης θα πρέπει να εργαστούμε και για τις μας προέλευσεις των εισαγόμενων προϊόντων. Μίλησαμε για την αμοιβαιότητα στι δημόσιε συμβάσεις, ε, δεν θα επανέλθω, αλλά είναι ένα μοχλός αυτός. Και επίση, ε, μαζί με μια πιο επιθετική πολιτική σε τομεί ε, έρευνας, καινοτομίας, τεχνολογίας, χρηματοδότησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρχει και μια καλύτερη αμυντική πολιτική σε όλε τι περιπτώσει που θα μπορούν να χρησιμοποιείται όταν χρειάζεται να έχουμε κάποιους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, εμείς καθυστερούμε πάρα πολύ να τα χρησιμοποιήσουμε, ενώ άλλες χώρες το κάνουν πιο γρήγορα. Δεν έχουμε ίσα όπλα λοιπόν. Και φυσικά όλα αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν και με το νομισματικό dumping. Υπάρχουν και τα θέματα της ανταγωνιστικότητας γενικά το πόσο βάρος έχει η ανταγωνιστικότητα, το χρόνο εργασία, όλα αυτά βαραίνουν και στην ευρωπαϊκή οικονομία και υπάρχει και ένα ζήτημα που θεωρώ πάρα πολύ ευαίσθητο και ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε και είναι το θέμα των προτύπων. Εμείς ε, ε, δεν ε, διστάζουμε να έχουμε πάρα πολύ δεσμευτικούς κανόνες σε όλους τους τομείς, στον τομέα της υγείας, του περιβάλλοντος, πολύ ωραία. Αλλά αυτοί οι κανόνες ε, στο διεθνή ανταγωνισμό μας φέρνουν σε δινή θέση ενίοτε. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό το θέμα, μήπως κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να προσθέτουμε κανόνες, μήπως θα πρέπει να επιβάλλουμε κανόνες στον εαυτό μας, θα πρέπει να το κάνουμε έτσι ώστε και τα προϊόντα που έρχομαι σε μέσα να σέβονται τους ίδιους κανόνες, ε, για να μην βρισκόμαστε σε κατάσταση ανισορροπίας. Αυτές είναι κάποιες ιδέες που θέτω επιτάπητος αλλά σήμερα δεν είναι πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι ζωτικό αυτό το ζήτημα της εκβιομηχάνησης της Ευρώπης και για την πραγματική βιομηχανική πολιτική. Πιστεύω ότι ήρθε ο χρόνος ε, να αποκτήσουμε τα μέσα και την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η Κομισιόν δεν ε, θα έχουν από μόνοι τους τα μέσα να το κάνουν, αλλά χρειάζεται κοινή πολιτική βούληση και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν σήμερα 27 βιομηχανικές πολιτικές και δεν υπάρχει μία πολιτική, βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ αυτό θεωρώ, Πρόεδρε, ότι πρέπει να συζητήσουμε και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σερνές. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Προύστ, θέλετε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλα σε υπόθηκαν ε, από την συγγήτρια και σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ. Πιστεύω ότι η βιομηχανική μας πολιτική συνδέεται με την εμπορική μας πολιτική και αντιστρόφως, ε, έχω πάρα πολλά ερωτήματα, δηλαδή να ξεκινήσουμε τον ορισμό του ίδιου του θέματος. Τι είναι μια ευρωπαϊκή επιχείρηση. Για μένα υπάρχουν τρεις πιθανές, τρεις δυνατές απαντήσεις. Μια ευρωπαϊκή επιχείρηση είναι καταρχήν μια επιχείρηση της οποίας η έδρα βρίσκεται στην Ευρώπη, ακόμη και αν έχει μονάδες παραγωγής σε μία περισσότερες τρίτες χώρες. Δεύτερον, ε, ε, ακόμη και αν μία μονάδα παραγωγή βρίσκεται στην Ευρώπη, αλλά η έδρα τρίτη χώρα. Και τρίτον, μία επιχείρηση τη οποία και η έδρα και οι μονάδε παραγωγή είναι στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται για τα τρία, αυτό το πρόβλημα ορισμού ε, πρέπει να το λύσουμε αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών ε, υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει τις μονάδες παραγωγής στην Κίνα. Έτσι λοιπόν ε, διακινδυνεύουν να πέσουν στην συνέπεια στο μέτρο αντι-dumping. Έτσι λοιπόν εδώ συνειδητοποιούμε ότι αν δεν έχουμε ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ε, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις μας, στις βιομηχανίες μας να πάρουν την σωστή απόφαση. Και για να έχουμε αποτελεσματική βιομηχανία θα πρέπει η εμπορική μας πολιτική να είναι διαρθρωμένη. Θα πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα και όχι κατακαιρματισμένη. Υπάρχει σήμερα μία κακή μεθοδολογία, ε, όμως ε, αυτή τη φορά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε την κατάσταση. Αν θέλουμε οι επιχειρήσεις μας να εξάγουν καλύτερα, θα πρέπει να υποφελούνται από ένα σαφές νομικό πλαίσιο που θα είναι ασφαλές και προβλέψιμο. Αλλά θα πρέπει επίσης οι αγορές των τρίτων χωρών να είναι ανοιχτές. Θα εξετάσουμε τρεις προτάσεις της Κομισιόν που θα έχουν καθοριστικές συνέπειες στις επιχειρήσεις μας. Η έκθεση του Ντανιέλ Κασπάρη που μας έχει απασχολήσει τα μάλα και ελπίζω να ολοκληρωθεί και συμφωνώ και με τη θέση της ηγήτρες όταν είπε σήμερα ε, ας θέσουμε αυτό το ζήτημα και σταματήσουμε να είμαστε ανόητοι θέλουμε εμείς ε, μια Ευρώπη που να δρέπει, έχουν και την έκθεση Ρινάλντι σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματο τη Ένωση για την εφαρμογή και το σεβασμό των κανόνων για το διεθνέ εμπόριο για μια πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά τον εξυγχρονισμό των μέσων εμπορική άμυνα που ελπίζουμε θα έρθει πριν το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να δούμε αυτά τα τρία μελλοντικά κείμενα ως σύνολο για να βελτιώσουν την πρόσβαση μας τρίτες χώρες και χωρίς αυτή την ε, συνοχή, τη μελλοντική, δεν θα προχωρήσουμε. Αυτή η ανάγκη συνοχής δεν θα πρέπει να σταματήσει τα τρία αυτά κείμενα. Πρέπει να υπάρχει και στις διμερείς μας ε, σχέσεις και πιο συγκεκριμένα όταν διαπραγματευόμαστε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών είναι λογικό σε κάθε διαπραγμάτευση να κάνουμε παραχωρήσεις. Δίχως ε, αυτό ποτέ δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε κανένα συμβασμό και να συνάψουμε καμία συμφωνία. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις ε, σε ε, χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι τελικά πουλάμε την ουσία του πλούτου μας. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η γνωμοδότηση θα μας χρησιμεύσει για να καθορίσουμε τα αμυντικά και τα επιθετικά συμφέροντα της βιομηχανίας μας, στο οποίο πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι. Και αναφέρθηκε και η Μαριέλ σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι τελευταίο που δεν πρέπει να ξεχνάμε και είναι πολύ σημαντικό. Είναι τα δικαιώματα διανοητική ιδιοκτησία. Είμαστε μια ήπειρο καινοτομία και πρέπει να προστατεύσουμε τους ε, εφευρέτες μας, διαφορετικά θα φύγουν. Αυτές οι προτάσει είχα να κάνω επιγραμμικά. Δεν θα μακρηγορήσω για να αφήσω χρόνο και στους υπόλοιπους συναδέλφους σας. Ευχαριστώ. Le prochain... Euh, Επόμενος ομιλητής, κύριος Λάγκε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος ε, Βέμπερ αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι με τον ε, πρόεδρο του να είναι εδώ. Θα μιλήσω εγώ στη θέση του. Εδώ και πάρα πολύ καιρό συζητούμε τους, ε, το βασικό προσανατολισμό τη βιομηχανική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση πριν από δύο χρόνια. Πέρυσι ε, ψηφίσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο και για ένα ψήφισμα και είναι ξεκάθαρο λοιπόν το πού θα προσανατολιστούμε και τι θέλουμε, πού θέλουμε να οδηγήσουμε την βιομηχανική μα πολιτική. Τώρα όμω, με την ανακοίνωση τη Επιτροπής είμαι κάπω απογοητευμένο, διότι γράφονται πολλά αλλά λείπουν τα μέτρα και πιστεύω ότι αυτό είναι ενδεικτικό στο ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς λέμε ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να έχει ως κέντρο της κήψη, την προτεραιότητα την εκβιομηχάνηση της Ευρώπης και όταν βλέπω πώς αντιδρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι προτάσεις υποβάλλει, τότε πιστεύω ότι δεν το πετυχαίνει αυτό, διότι πάντα βρίσκουμε προτάσεις οι οποίες αντιβαίνουν στα συμφέροντα της ε, βιομηχανίας μας, ε, είτε στον τομέα της ανανταγωνιστικότητας, ε, είτε ορισμένες φορές στην ενιαία αγορά και πιστεύω ότι εδώ πραγματικά πρέπει να θέσουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες έτσι ώστε πραγματικά η βιομηχανική πολιτική να βρίσκεται στο κέντρο της πολιτική μα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακαλώ την Επιτροπή να αντιδράσει με συνέπεια και συνεκτικότητα. Και εδώ να τονίσω και να συμφωνήσω με αυτό που είπε η συγγήτρια, ότι αυτό θα γίνει σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ήδη έχουμε ζητήσει το, να ανανεωθεί να χρησιμοποιηθεί το άρθρο 179. Έχει τις γενικές κατευθυντήριε γραμμές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική και μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου. Και όταν βλέπω σε επιμέρους, τους επιμέρους τομείς, στον τομέα του εμπορίου, ε, παρατηρώ, να σας πω ότι το εμπόριο δεν είναι αυτός σκοπός με το εμπόριο. Θέλουμε να προωθήσουμε τα ε, βιομηχανικά μας, τα βιομηχανικά μας συμφέροντα και αυτό θα δώσει και αποχρώσεις στην πολιτική μας. Ελπίζω πραγματικά να το καταφέρουμε στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών καλύτερα, διότι φυσικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχουν άλλα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ε, ε, στον τομέα των ε, μηχανικών κατασκευών, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην, στον τομέα της χημικής βιομηχανίας. Εκεί πέρα υπάρχουν ξεκάθαρα πρότυπα, εκεί πέρα υπάρχουν ξεκάθαρες εφορολογικές απόψεις, προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά και αυτά τα συμφέροντα ακολουθούνται και εμείς εδώ πραγματικά θέλουμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας μας, τις δουλειές και την βιομηχανία μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Ντεσάν μας ε, ανέφερε διεξοδικότατα τις ε, λεπτομέρειες στην έκθεσή της και να την συγχαρώ. Καταρχάς συμφορώ με, τις, ε, με τα δάνεια και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πιστεύω πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να προωθήσουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύω ότι η συγκέντρωση των ερευνητικών μας δυνατοτήτων είναι κάτι που πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουμε. Το μόνο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά ακόμα από το στόχο της αγοράς και θα χρειαστούμε και οικονομική βοήθεια στην, ε, να δοθεί στην έρευνα διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι εταιρείε ε, διαφυλάσσουν με, κάθε μέσο τις, ε, τα αποτελέσματα των δικών τους ερευνών. Δεν θέλουν να τα μοιράζονται. Τώρα, να πω ότι αρχίζω και ανησυχώ όταν αρχίζουν να γίνεται λόγος για προστασία και ε, μηχανισμούς άμυνας του, και προστασία του εμπορίου, διότι η άμυνα σημαίνει και μια επίθεση και θα σου γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Και πιστεύω ότι σωστά πρέπει να εστιάσουμε στην ε, τωρινή κατάσταση της οικονομίας με τις απώλειες των θέσεων εργασίας, κάτι καταστροφικό από πολλές απόψεις. Έχει πλήξει και την, ε, βιομηχανία, τον, ε, την κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη δεν πιστεύω, ότι πρέπει να, ε, δεν πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε με όλα, αλλά να έχουμε υπόψη λίγα πράγματα. Εγώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της ε, κατασκευαστικής βιομηχανίας και το τα ωφέλη που έχουμε αποκομίσει από αυτήν και να δούμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε το κέρδος. Έπειτα, για το χρονικό διάστημα μέχρι 30 ετών, πιστεύω πως πρέπει να κοιτάξουμε όσο το δυνατόν πιο στο μέλλον γίνεται και να δούμε τι γίνεται και με τον δευτερογενή τομέα, διότι οι πρώτες πιστεύω ότι όπως είπε και η συγγήτρια ε, υπάρχει, έχουν κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε και να διαμορφώσουμε δράσεις οι οποίες θα αποτρέψουν το αρνητικό αντίκτυπο και θα δώσουν ίσους όρους σε όλους. Επίσης, χρειαζόμαστε νέε νέες συμφωνίες, χρειαζόμαστε περισσότερη προσοχή ε, και χρηματοδότηση στην έρευνα, στην ε, βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, ίσως ε, βελτίωση των όσων ήδη κάνουμε. Και αυτά είναι, αυτή είναι για τους οποίους πραγματικά πιστεύω πως πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή. Και σας ευχαριστώ ξανά, εισηγήτρια, για την εξαιρετική σας έκθεση. Ευχαριστώ τη Μαρία Λτεσταρνές για την παρουσίαση που κάνει και για τους στόχους, τους φιλόδοξους που θέτει όσον αφορά τη βιομηχανική πολιτική. Έχει δίκιο ο Μπέντ. Έχουμε ξεκινήσει εμπορικές διαπραγματεύσεις με όλες τις περιοχές του κόσμου. Πολλές φορές όμως δεν ξέρουμε τι ακριβώς ζητάμε για τη βιομηχανία μας επί χρόνια η Επιτροπή θεωρούσε ότι μία οικονομία που βασίζεται στις υπηρεσίες αρκεί για να εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες των Ευρωπαίων. Ευτυχώς, σήμερα ξεκινήσαμε μία συζήτηση για το θέμα της βιομηχανίας στην Ευρώπη και θα σας πω σαν παράδειγμα ότι πριν από τρεις εβδομάδες με κάποια μέλη του Κοινοβουλίου οι οποίοι εμπλέκονται και στην έκθεση επί τους ουσίας, στην οποία αναφέρεται αυτή η γνωμοδότηση, συναντήσαμε τους ε, επικεφαλείς του ομίλου Αρσελόρ Μιτάλ, οι οποίοι μας μίλησαν για τις ε, δωρεάν ποσοστώσεις που ζητούν. Έχουν πάνω από δύο δις σήμερα. Ε. Μας ζητούν αυτές τις δωρεάν ποσοστώσεις μέχρι το 2020-2030. Ο Επίτροπος Ταγιάννη πρότεινε κάτι, ευτυχώς κάποιος τον διόρθωσε, πρότεινε να χρηματοδοτήσει ο προϋπολογισμός ο ευρωπαϊκός τον όμιλο Μιτάλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι σήμερα σε όλα τα κράτη υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση του ομίλου αυτού. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είδατε εργαζόμενους από όλη την Ευρώπη που εργάζονται στον όμιλο αυτό, οι οποίοι ήρθαν για να μας πούν ότι μια χαλιβουργία η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη στην Ευρώπη είναι μια χαλιβουργία που λειτουργεί με εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, που παράγει χάλιβα που χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες με υψηλή προστιθέμενη αξία και σε κάθε περίπτωση ο ανταγωνισμός στον οποίο αναφερόμαστε στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ανταγωνισμός που αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων, αλλά αποκλειστικά και μόνο τις τεχνολογίες, την καινοτομία και ακριβώς αυτό πρέπει να βάλουμε στην καρδιά της συζήτησής μας. Το ίδιο είπαμε και για τον άνθρακα. Στην Επιτροπή καταψηφίσαμε την αποτελεσματικότητα του άνθρακα. Γιατί? Γιατί η πολιτική μας είναι να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και όχι να τις οδηγήσουμε προς ένα μελλοντικό προσανατολισμό. Σκοπός μας στην Ευρώπη είναι όχι να στηρίξουμε τις νέες τεχνολογίες και το μέλλον των επιχειρήσεών μας, αλλά να βοηθήσουμε την εγκατάλειψη από μέρους των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων της Ευρώπης. Το βλέπουμε σε όλους τους τομείς και στην ε, προσέγγιση που έχουμε, παραδείγματος χάρη, και για τον τομέα της αεροναυτιλίας. Βλέπουμε ότι ισχύει η ελάχιστη ρύθμιση, κάτι που οδηγεί στις τις επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν την Ευρώπη. Τώρα, όταν αναφερόμαστε στον εμπορικό τομέα και είδαμε ότι σαφώς και οι διάφορες διατάξεις θα πρέπει να στηρίζουν και να ευνοούν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να είναι σαφές το κείμενο της οδηγίας όσον αφορά την προστασία, γιατί πραγματικά αυτό πρέπει να κάνουμε, να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας σε σχέση με ξένες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της ΓΚΟΕ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα που συζητούμε σήμερα και θα συζητήσουμε το Γιάννικ ότι είναι θύματα οι εργαζόμενοι στον όμιλο Αρσελόρ Μιτάλ, θύματα της παγκοσμιοποίησης. Και βλέπουμε ότι αυτό συμβαίνει σε πολλούς τομείς στην Ευρώπη. Για την δική τους περίπτωση είναι σαφές αυτό που γίνεται. Υπάρχει μια ανταγωνιστική επιχείρηση βιώσιμη και εδώ βλέπουμε ότι η στάση της ε, Γαλλίας παραδείγματος χάρη έναντι αυτών των εργαζομένων είναι κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμείς εδώ να το στηρίξουμε. Και πρόκειται απλώς για ένα παράδειγμα αυτών που λέμε. Είναι κάτι που ξεπερνάει αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση γιατί εδώ έχουμε 26 εκατομμύρια ανέργους σε όλη την Ευρώπη. Και το ερώτημα είναι γιατί η Ευρώπη χάνει τη βιομηχανία της. Υπάρχουν πολλές εξηγήσει, αλλά ένας καθοριστικός παράγοντας είναι η τρομερή μείωση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη. Και η εταιρεία συμβούλων McKinsey, η οποία πέρσι έκανε μία μελέτη για το θέμα αυτό και για τις νέες προκλήσεις, ανέφερε ακριβώς αυτό το παράγοντα μεταξύ του 2007 και 2011 μειώθηκαν οι επενδύσεις τέσσερις φορές παραπάνω από τη μείωση του ΕΕΠ στην ίδια περίοδο. Αναφέρομαι στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Επαναλαμβάνω, ε, τέσσερις φορές περισσότερη μείωση από αυτή της πτώσης του ΕΕΠ και 20 φορές παραπάνω περισσότερη μείωση, 20 πλάσια μείωση σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης την ίδια περίοδο 2007-2011. Οι επενδύσεις λοιπόν μειώνονται και αυτό οδηγεί στην ραγδαία μείωση της βιομηχανικής δραστηριότητας. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι 750 δις είναι τα πλεονάσματα των επιχειρήσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό τα αποθέματα ε, ρευστότητας μεταξύ 2007 και 2011 δεν επενδύθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Και ο καπιταλισμός στον δυτικό κόσμο, στην Αμερική, στη Δυτική Ευρώπη, οδηγεί σήμερα σε μια πολύ σημαντική μείωση των επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ των ίδιων χωρών. Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι ότι το σχέδιο της Επιτροπής να δώσει κίνητρα για περισσότερες επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα δεν πρόκειται να φέρει αποτελέσματα, καθότι αυτό που αναφέρουν σαν κίνητρο δεν πρόκειται να οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις. Είδαμε ότι τα κέρδη αυξάνονται και το αντίστοιχο ποσοστό επενδύσεων, η ρευστότητα δηλαδή που επανεπενδύεται στον τομέα αυτόν, μειώνεται. Και υπάρχουν δισεκατομμύρια ρευστότητας, δισεκατομμύρια τα οποία δεν επενδύονται στη βιομηχανία και την ίδια ώρα 26 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω λοιπόν, η λύση δεν πρόκειται να είναι αυτή που περιμένουμε με αυτά τα κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσουμε ομίλους σαν την ArcelorMittal στην επένδυση στον τομέα αυτό. Τους δώσαμε κίνητρα. Παρόλα αυτά δεν θέλουν να επενδύσουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλου είδους μέτρα χρειαζόμαστε άλλου είδους επενδύσεις που δεν προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά από τον δημόσιο και αυτό έτσι ώστε να υπάρξει πραγματικός δημοκρατικός έλεγχος των εργαζομένων επί των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Πρέπει να βάλω κάποια όρια χρόνου, γιατί μας έχουν μείνει μόνο 10 λεπτά για αυτό το θέμα και θέλουμε να ακούσουμε και την Κομισιόν και την εισηγήτρια. Δύο άτομα έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο, κύριε Πίτερ. Τρία λεπτά. Θα είμαι πολύ σύντομη. Είναι ενδιαφέρον ε, που βλέπουμε την ε, βιώσιμη εκβιομηχάνηση. Φαίνεται σαν οξύμορο. Ο όρος ε, εκβιομηχάνηση φέρνει μνήμες βαριές βιομηχανίας. Και παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι είναι βιώσιμο στο μέλλον και επομένω, ε, είναι δύσκολο να φανταστούμε αυτό το συνδυασμό. Νομίζω ότι η Μαρία Ελή είπε πολλά, ένα ολόκληρο κατάλογο από πράγματα που πρέπει να κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα προς το μέλλον, ε, να έχουμε ευέλικτη χρηματοδότηση, προστασία διανοητικών δικαιωμάτων, και υπάρχουν πάρα πολλοί καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότηση που αναδύονται και πρέπει να έχουμε ευέλικτο τρόπο σκέψη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα απορρίθμιση, αλλά πρέπει να σκεφτούμε έξω από το κουτάκι. Επίσης, πρέπει να δούμε πώς θα σώσουμε κάποιες αποτυχημένες ε, επιχειρήσεις. Ε, γιατί ξοδεύουμε χρόνο να σώζουμε εγχειρήματα του παρελθόντος. Υπήρξε στο παρελθόν ε, ανησυχία για την ε, πληθυσμιακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα της Ευρώπης ε, και σκεφτόμασταν ε, τι θα κάναμε τότε, αλλά κανείς ε, δεν είχε σκεφτεί να αναγνωρίσει ότι θα έρχονταν και τα αυτοκίνητα και τα αυτοκίνητα έφεραν την αλλαγή που κανείς δεν είχε προβλέψει. Έτσι λοιπόν, αν δούμε το μέλλον, πρέπει να δούμε τι υπάρχει εκεί. Οι δομές λοιπόν που θα συστήσουμε θα πρέπει να είναι ευέλικτες και να μπορούν να συνδυαστούν με καινοτομίες που δεν έχουμε καν σκεφτεί ότι είναι δυνατόν να συμβούν. Τα τελευταία 5-10 χρόνια έχουμε διαφορετικό εξοπλισμό στα χέρια μας. Δεν θα έχουμε σκεφτεί αυτό πριν δεκαετή. Και έρχομαι στο τελευταία παρατήρησή μου. Ακούσαμε για την έρευνα και πόσο ζωτική σημασία είναι, αλλά θα πρέπει να ασκούμε επίση και για την παιδεία. Δεν ε, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα σκέφτονται μέσα στο κουτί, θέλουμε ανθρώπους που θα σκέφτονται έξω από το κουτί, γι' αυτό θέλουμε να τους καταρτήσουμε, να είναι ικανοί πολίτες της Ευρώπης, να μπορούν να προσαρμοστούν. Ξέρουμε ότι αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή, αυξάνεται η στάθμη της ε, θάλασσας, το θέμα της επιστημικής ασφάλειας. Ε, όλα αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και χρειαζόμαστε ένα εργατικό δυναμικό που να μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις προκλήσεις. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Dartmouth. Είναι πραγματικά εκφοβιστικό να μιλά κανείς ε, μετά από τους κύριους Μέρφη και Ζαντό, γιατί είναι πολύ γλαφυροί Λοιπόν, για την ε, βιομηχανία θα ζητήσω από τους συναδέλφους να σκεφτούν τα αποτελέσματα της ενεργής πολιτικής για την αποβιομηχάνηση. Αν καταστήσετε την ενέργεια πιο ακριβή, μία από τις συνέπειες αναπόφευκτα θα είναι η αποβιομηχάνηση. Παραδείγματος χάρη στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε ε, τρία ε, εργοστάσια ε, αλουμινίου που έπρεπε να κλείσουν γιατί η ενέργεια ήταν πολύ ακριβή. Γιατί οι ευρωπαϊκές πολιτικές που τις, τις έχουν εμπνευστεί οι πράσινοι και η γκουε και πάντοτε είναι πολύ αποτελεσματική πολιτική. Το λέω εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Συγγνώμη, αλλά δεν έδωσα το λόγο σε εσά, κύριε Ζαντό. Σα ε, επενώ για <laughs> τι δεξιότητε, σα ω πολιτικό και για την κλαφερότητά Σα Δεν μπορείτε να περιμένετε να συμφωνώ και μαζί σα για το θέμα της διαφάνειας ε, και το θέμα της διαφάνειας της Κομισιόν μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό. Και θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους και από τα κόμματα που εκπροσωπούν και από τους φιλελευθέρους ε, να σκεφτούν τα αποτελέσματα ε, των πολιτικών τους για την ενέργεια, για τις θέσεις εργασίας, για την ανάπτυξη και για την αποβιομηχάνηση σας. Ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε την Επιτροπή. Ο κύριος Μάρτιν. Ναι. Δεν είμαι ο κύριος Μάρτιν. Συγγνώμη, είχα δύο ονόματα, δεν ήξερα ποιος είστε. Καλό σας βράδυ. Και σας ευχαριστώ που μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο για να εξηγήσω αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχει μία νέα μορφή. Εμείς δεν αλλάζουμε κάτι σε σχέση με τους ε, στόχους του 2010. Απλώς θεωρήσαμε ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση τόσο που εδώ χρειάζεται ίσως να κινητοποιήσουμε λίγο την βιομηχανική μας πολιτική και να την αλλάξουμε λίγο. Αυτό που προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε με αυτήν την ε, ανακοίνωση είναι κάτι από αυτά που ακούστηκαν. Πρώτον, να συνεχιστούν οι επενδύσεις. Και χτες και σήμερα σε κάποια άλλα βήματα είπα αυτά που λέει και η έκθεση McKinsey. Πώς μπορούμε λοιπόν να κινητοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις. Είτε να αντικαταστήσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις με δημόσιες επενδύσεις, αλλά στην ίδια έκθεση λέει ότι μόνο 2% αν θέλετε είναι το ύψος των επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μαζί. Και σε κανονικές περιπτώσεις αυτό το ποσοστό φτάνει το 20%. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να έχουμε αποτελέσματα. Πρώτον, κάτι που ήδη έχει κάνει η Επιτροπή, να εντοπίσει δηλαδή έξι τομείς που να έχουν ραγδαία ανάπτυξη βάσει κινέζικων, ιαπωνέζικων, βρετανικών και αμερικανικών εκθέσεων με διπλάσιους ε, ρυθμούς ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για τομείς και δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας, προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε τα επόμενα δύο ή τρία χρόνια να δημιουργηθούν πρότυπα για να αναπτυχθούν αυτοί οι τομείς και να δημιουργηθούν οι συνθήκες αυτές στην αγορά που θα οδηγήσουν σε καινοτομία, όπως παραδείγματος χάρη για τις ε, περιπτώσεις ανάπτυξης της αγοράς των έξυπνων δικτύων, μέτρα τα οποία βεβαίως δεν αρκούν. Θέλουμε να δώσουμε κίνητρα στις επενδύσεις, κάτι που προϋποθέτει πρώτον τη δημιουργία συνθήκων για τις αγορές και δεύτερον κάτι που ήδη έχει ξεκινήσει, που έχει προβλεφθεί για τις εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές, που είναι καλύτερη προστασία των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όπως παραδείγματο χάρη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ενδιάμεσες ε, επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δηλαδή μέσου μεγέθους, οι οποίες καλούνται σήμερα να ανταγωνιστούν ε, στις αγορές άλλων χωρών με πολύ διαφορετικές συνθήκες. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι όσον αφορά την παραγωγική επένδυση στην Ευρώπη, η επιλογή ε, πολλές φορές καθορίζεται από το επίπεδο προστασίας που παρέχουμε στις επιχειρήσεις. Επίσης, ο Επίτροπος Ταγιάννη ξεκίνησε την Mission for Growth, αποστολή για ανάπτυξη, κάτι που άμεσα θα οδηγήσει όχι μόνο στο άνοιγμα των αγορών, αλλά και στην πρόσβαση στις πρώτες ύλες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τις ε, προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Συμπεριλαμβάνουμε λοιπόν στα μέτρα προώθησης ε, το θέμα των δεξιοτήτων και προσόντων για τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα έχουν αποτέλεσμα. Η ανακοίνωση αυτή είναι απλώς το πρώτο βήμα σε μία σειρά μέτρων που καλούμεθα να υιοθετήσουμε. Γι' αυτό και όλοι οι εμπλικόμενοι φορείς θα πρέπει να μας στηρίξουν, να συνεργαστούν. Ελπίζουμε ότι θα είναι αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα. Αλλά βεβαίως πολλές τέτοιες ανακοινώσεις έγιναν στο παρελθόν χωρίς να έχουν το έβρος της σημερινής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια έχει το λόγο για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω στην Επιτροπή ότι βεβαίως συμφωνώ με το πνεύμα της πρότασής σας. Περισσότερη βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά όμως θα ήθελα να πω ότι όταν ακούω την Επιτροπή που λέει ότι διαλέγω έξι τομεί που θα είναι οι τομείς ανάπτυξης, διψήφιας ανάπτυξης, εγώ δεν ξέρω βάσει ποιων κριτηρίων αποφασίζει η Επιτροπή για το ποιε θα είναι οι μελλοντικέ δυνατότητε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και σε καμία περίπτωση μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Η ανάπτυξη κυρίως προέρχεται από υψηλή τεχνολογία, από τις επιχειρήσεις, από τους δημιουργούς, από τους ε, τεχνικούς, αλλά όχι από την Επιτροπή. Διαφωνώ λοιπόν και το λέω για να είμαστε σαφείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούν τα κράτη-μέλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε κάποιους ε, στρατηγικούς τομείς. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στη θέση των επιχειρήσεων. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε, να τους στηρίξουμε, να τους ευνοήσουμε, να τους δώσουμε κίνητρα όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αλλά ε, βλέπω ότι διαφωνείτε και εγώ διαφωνώ μαζί σας. Δεν είναι δυνατόν εμείς να αποφασίσουμε για το ποιοι είναι οι τομείς στρατηγική σημασία και ανάπτυξη για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν του συναδέλφου. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε εδώ. Ακούστηκαν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους Κιώδες και τους άλλους και ε, θεωρώ ότι συμφωνούμε μεταξύ μας η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ενισχυθεί όσον αφορά την ε, βιομηχανική πολιτική, καθότι δεν μπορούν αυτά να γίνουν χωρίς ε, τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Συμφωνήσατε όλοι ότι χρειάζεται περισσότερη συνοχή στην εμπορική μας πολιτική, ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα για την προστασία Μιλήσατε για ένα σαφές νομικό πλαίσιο, το οποίο δεν θα αλλάζει μεσοπρόθεσμα. Κανείς δεν μπορεί να επενδύσει αν δεν υπάρχει σταθερότητα για τις επενδύσεις και νομική ασφάλεια. Είπατε επίσης ότι η προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη πρέπει να βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία, στην καινοτομία και στην εξοικονόμηση των πόρων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσον αφορά τις αποδοχές των εργαζομένων μας. Η καλύτερη αν θέλετε, η οικονομική ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός της Ευρώπης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βασιστεί σε χαμηλότερες αποδοχές, ανταγωνιστικές αποδοχές. Ο προϋπολογισμός για την έρευνα, εδώ θα πρέπει να καθοριστούν κοινοί στόχοι και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να λειτουργήσουν συλλογικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση αυτού του προϋπολογισμού για την έρευνα στην Ευρώπη. Είμαστε μπροστά όσον αφορά την καινοτομία και σαφώς και η επένδυση στην κατάρτιση και στις δεξιότητες των Ευρωπαίων εργαζομένων είναι κάτι το οποίο σήμερα είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο θα πρέπει να διατηρήσουμε. Τα πνευματικά δικαιώματα επίσης είναι κάτι που θα πρέπει να το προστατεύσουμε. Αυτά Μπορείτε να ολοκληρώσετε παρακαλώ, λέει ο Πρόεδρος. Επόμενο σημείο. Μάλλον όχι, προθεσμία 26 Απριλίου λοιπόν. Για το σχέδιο έκθεσης θα παρουσιαστεί τότε από τον εισηγητή μας. Επόμενο και τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα παριθμών 12, ενδιάμεση συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέση, Ευρωπαϊκή Κοινότητα και Κεντρικής Αφρικής. Εισηγητής ο Ντέιβιντ Μάρτιν, είναι μία διαδικασία συνένεση, είναι μία από τι συμφωνίε Αφρική, ε, των ομάδων Αφρικής ΑΚΕ. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Και σήμερα Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους από το Καμερούν, την, τον πρέσβη Ντάνιελ Εμπίν Αβί, με ένα μέλος της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Συνέλευσης του Καμερούν, Γιώζεφ Ονκόνο, και τέλος ένας ε, αντιπρόσωπος ε, τον συνδέσμων, επαγγελματικών συνδέσμων του Καμερούν, Εμπάρκα Ατανγκάνα. Αυτοί οι καλεσμένοι παρευρίσκονται και πιστεύω η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως γνωρίζετε τώρα δρομολογούνται αρκετές συμφωνίες με το Καμερούν και φυσικά με την ε, περιοχή της Κεντρικής Αφρικής συνολικά. Ωστόσο, μια το, και το Καμερούν είναι η μόνη κεντροαφρικανική χώρα που έχει υπογράψει την ενδιάμεση συμφωνία και επειδή το Καμερούν είναι η μεγαλύτερη και δυνατότερη οικονομία της περιοχής, έχει μια ιδιαίτερη και πολύ σημαντική θέση στην ε, οικονομία της περιοχής και στην ε, διαδικασία ολοκλήρωσης της περιοχής αυτής. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό που ήρθαν σήμερα αντιπρόσωποι του Καμερούν στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής. Ας αρχίσουμε με τον David Μάρτιν, τον εισηγητή της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου τους εκλεκτούς μας καλεσμένους από το Καμερούν. Έχετε απόλυτο δίκιο είναι πολύ σημαντική χώρα, ζωτική σημασία χώρα στην κεντροαφρικανική περιοχή. Ε, έγιναν διαπραγματεύσεις 25 Ιανουαρίου του 2009. Μας πήρε μόνο τέσσερα χρόνια μέχρι να το λάβουμε. Τι λάβουμε από το Συμβούλιο, τελικά τι λάβαμε όμως. Και επειδή εμείς είμαστε γρήγοροι, γίνονται και γρήγορα οι διαδικασίες. Γιατί αν περιμέναμε <laughs> από το Συμβούλιο θα ακούσαμε και περισσότερο. Ε, εμείς το θεωρούμε ένα ακόμα λιθαράκι παρά μια ενδιάμεση συμφωνία. Και να σας πω την αλήθεια, μου αρέσει και αυτή η διατύπωση, διότι πιστεύω πως ταιριάζει περισσότερο. Είναι κάτι ανάμεσα στην ενδιάμεση συμφωνία και στην ολοκλήρωση των ε, τη Συμφωνία Οικονομική Εταιρική Σχέση, όχι μόνο με το Καμερούν, αλλά και με γενικότερα την Κεντρική Αφρική. Σε γενικέ γραμμέ πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό επίτευγμα και για το Καμερούν και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την βελτίωση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στους ε, δύο. Και πιστεύω ότι οι σχέσεις αυτές θα βελτιωθούν ε, σημαντικά λόγω της συμφωνίας αυτής. Ε, υπάρχει πρόσβαση ελεύθερη από δασμούς από προϊόντα του Καμερούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό πιστεύω είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ανοίξει σταδιακά η αγορά του Καμερούν στους, ε, για τους παραγωγούς. Όσον αφορά τις αναπτυξιακές ε, πτυχές, η συμφωνία αυτή αντιμετωπίζει τα ζητήματα, για παράδειγμα, των τεχνικών ε, φραγμών στο εμπόριο και της επίλυσης των διαφορών όπως σας είπα, είναι ένα ακόμα λιθαράκι προς την ολοκλήρωση και φυσικά οι συζητήσεις θα συνεχιστούν, ιδιαίτερα όσον αφορά την επισήμανση προέλευσης, τις υπηρεσίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καλή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου. Και το τελευταίο αυτό, το κράτος δικαίου, μας θα υπενθυμίζει το καθήκον μας να βοηθήσουμε το Καμερούν δεδομένης και της απαγωγής εχθές στο Καμερούν 7 Γάλλων ε, υπηκών Πιστεύω λοιπόν πως θα επωφεληθούμε αμοιβαία από αυτή την συμφωνία. Το Καμερούν ε, βελτιώνει το κράτος δικαίου του και προστατεύει τους δικούς μας πολίτες. Τώρα όσον αφορά την ολοκλήρωση που είναι και το πιο σημαντικό και βαθύτερο ζήτημα, εκεί ε, διαπραγματευόμαστε μόνο με το Καμερούν και όχι με την Κεντρική Αφρική. Δυστυχώς. Και δυστυχώς διότι το, να σας πω το Καμερούν αντιπροσωπεύει ένα τέταρτο των εμπορικών συναλλαγών μας με την ε, Κεντρική Αφρική και οι περισσότερες ε, άλλες ε, χώρες της περιοχής είναι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, έτσι κατατάσσονται και δυστυχώς δεν μπορούν να επωφεληθούν προς το παρόν από τις εμπορικές συναλλαγές μαζί μας. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που πρέπει να επιληθούν εκεί. Αλλά πιστεύω πως ε, η συμφωνία αυτή με το Καμερούν είναι ένα σημαντικό βήμα και πιστεύω, ελπίζω και πιστεύω εμείς και το Καμερούν να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να καταφέρουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη συμφωνία. Όμως ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος και αυτό, γι' αυτό θα σταματήσω και περιμένω να ακούσω από τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Ευχαριστώ πολύ. Ας τους ακούσουμε λοιπόν τον πρέσβη του Καμερούν, Ντανιέλ Εβινά Αμπέ Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι ο κύριος ε, Μάρτιν ε, περίγραψε συνολικά τη συμφωνία. Απλά ε, θα κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Πρέπει να πω από την αρχή ότι το Καμερούν χρειάζεται αυτή τη συμφωνία. Την υπογράψαμε. Εμείς έχουμε λοιπόν συμφέρον και Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, τη συμφωνία για να μπορούμε να συνεργαστούμε με την ευρωπαϊκή αγορά. Όμως, επίσης, ε, έχουμε έναν ε, ρόλο σε επίπεδο της Κεντρικής Αφρικής, τον οποίο πρέπει να παίξουμε, γιατί ο τελικός στόχος των συμφωνίων αυτών είναι η περιφερειακή ολοκλήρωση. Αυτή η ολοκλήρωση όταν υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία, μας αναγκάσαν να μην είμαστε λέγγυοι με τα σε άλλες χώρες της ε, Κεντρικής Αφρικής. Μας θεώρησαν ότι ήμασταν οι προδότες ε, για την περιοχή και οι άλλες χώρες ουσιαστικά είχαν τελείως διαφορετική ε, στάση. Αυτό είναι αλήθεια. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι με τις επιφυλάξεις οι οποίες ακούστηκαν από τους άλλους εταίρους μας στην Κεντρική Αφρική και όσον αφορά τα όσα έχουν αποφασιστεί, τελικά είδαμε ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε προς μια πιο γενική συμφωνία που να καλύπτει όλη την περιοχή. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα λέμε να προχωρήσουμε. Έχουν ξεκινήσει διάφορες προσπάθειες για να προσαρμοστεί το κείμενο και νομίζω ότι η ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα θα μου επιτρέψει να σας πω ότι ναι μεν το Καμερούν έχει υπογράψει, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει έτσι ώστε οι άλλοι αφρικανικοί εταίροι επίσης να πλησιάσουν το κείμενο. Μιλήσατε για τις οκτώ χώρες και οι υπόλοιποι, οι οποίοι βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, αν θέλετε, με εμάς αναπτυξιακό. Γιατί δεν έχει κυρωθεί ακόμα η συμφωνία. Διότι θεωρούμε ότι δεν είναι πλήρης η συμφωνία αυτή και γιατί θεωρούμε επίσης ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το πού βρισκόμαστε και τι κάνουν οι υπόλοιποι στην Κεντρική Αφρική. Θέλουμε λοιπόν να διαπραγματευτούμε, είμαστε διατεθειμένοι να διαπραγματευτούμε, αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να συμφωνήσει και η άλλη πλευρά. Και χρειάζονται υποχωρήσεις από τις δύο πλευρές, όπως είπε και κάποιος ε, βουλευτής πριν από λίγο και εδώ νομίζω ότι ομιλώ εξ ονόματος όλων των άλλων κρατών της περιοχής, πρέπει να προχωρήσουμε και η μεν και η δε. Από ό,τι ξέρω και δεν παρακολουθώ εγώ την υπόθεση, μου είπαν ότι δεν μας έχουν δοθεί όλα τα στοιχεία που ζητήσαμε από τους άλλους εταίρους στη διαπραγμάτευση. Περιμένουμε λοιπόν να μας βοηθήσετε έτσι ώστε να μας ακολουθήσουν και οι άλλοι αφρικανικοί εταίροι και να εξελιχθούν τα πράγματα όπως όλοι επιθυμούμε. Επιπλέον, ίσως δεν πρέπει να το πω αυτό εδώ, μας δόθηκαν κάποιες ελπίδες, οι οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Είναι εδώ κάποιοι αρμόδιοι για το θέμα της παραγωγής ε, μπανάνας, καλλιέργειας μπανάνας. Ξέρετε ότι από το 2009 περιμένουμε κάποια πράγματα που μας είχατε υποσχεθεί, έχει υπογραφεί συμφωνία και η συμφωνία αυτή δεν έχει υλοποιηθεί. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μας οδηγούν σε μια δυσπιστία και είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα και στις δύο επιτροπές που διαπραγματευόμαστε και στη ΣΕΜΑ και στην ΑΣΕ υπάρχουν κάποιες αλλαγές, κάποια πρόοδος και ελπίζω ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι η νέα ομάδα διαπραγμάτευσης έχει δεσμευθεί έτσι ώστε να προοδεύσουν οι διαπραγματεύσεις και αυτό το λέω και επαναλαμβάνω ότι πρέπει οι υποχωρήσεις να γίνουν και από τις δύο πλευρές και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε πεδίο για περισσότερη συνεννόηση. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Πρέπει να βάλουμε κάποια όρια χρονικά στους ομιλητές γιατί έχουμε λιγότερα από 15 λεπτά στη διάθεσή μας και πρέπει να ακούσουμε και κάποιους ομιλητές που έχουν δει στο λόγο. Ο κύριος Μέρφυ καταρχήν γιατί ήταν ο πρώτος που ζήτησε το λόγο. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω. Έξτρα 10 παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Ντεβίτ και τον ε, κύριο Πρέσβη κάποιες παρατηρήσεις. Ε, καταρχήν ε, ότι δεν ε, θα πρέπει να λέμε ότι οι συμφωνίες αυτές έχουν να κάνουν με περιφερειακή ολοκλήρωση γιατί τι και απαντάει η Κομισιόν στην κατάσταση αυτή όταν ε, δεν υπογράφουν τη συμφωνία και δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο κύριος Πρέσβη, αλλά έχει γίνει αξιολόγηση για τον αντίκτυπο των ε, συμφωνιών εταιρικής σχέση ε, στα έσοδα του από του δασμού, από τη στιγμή που εφαρμόζονται και στον αντίκτυπο της μεταπητική βιομηχανίας στο Καμερούν. Τρία, κατάλαβα ότι είπε ε, ο πρεσβευτή ότι θέλει το Καμερούν αυτή τη συμφωνία, αλλά θέλει περισσότερο πρόσβαση στι ευρωπαϊκέ αγορέ, Φυσικά το κατανοώ και συμφωνώ. Αλλά αν υπήρχε ένα άλλο τρόπο να έχετε πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, αν δεν χρησιμοποιούσε αυτό η Κομισιόν ε, ως ε, το καρότο ε, για τη χώρα σα, τότε τι θα επιλέγατε και έγιναν και δύο σχόλια για τις διαπραγματεύσεις ε, που ήταν ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να φερθείτε λεπτομερέστερα σε σχέση με τη στάση της Κομισιόν στι διαπραγματεύσει, γιατί ακούμε δύο πολύ διαφορετικέ ιστορίε. Μία από την Κομισιόν, ότι είναι πάρα πολύ ευέλικτη και διαθέσιμη να συζητήσει τα πάντα, αλλά εδώ ακούμε και μια άλλη ιστορία ότι δεν ισχύει πάντοτε κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα μα ενδιαφέρει να ακούσουμε λεπτομέρειε από αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όλα από όλοι για την περιφερειακή ολοκλήρωση. Δεν μακρηγορώ λοιπόν. Αν κατάλαβα καλά, η κύρωση επίσης έχει παγώσει μέχρι ολόκληρη η περιφέρεια να συμφωνήσει με την Κομισιόν. Μπορεί κάποιος να το επιβεβαιώσει αυτό. Και επίσης ε, να μας εξηγήσετε ποιες δυσκολίες βλέπει το Καμερούν και οι άλλες χώρες Κεντρικής Αφρικής με την υπογραφή της EPA. Θέλω επίσης να ρωτήσω τον πρέσβη ποιος βλέπει να είναι ο αντίκτυπος ε, στην ε, περιφερική ολοκλήρωση. Επίση, ακούσαμε ότι ο λόγος που έχει παγώσει ο κ. στο Καμερούν είναι επειδή υπάρχουν ε, διαφορετικές θέσεις σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Καμερούν. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε ποια μορφή λαμβάνουν οι θέσεις αυτές πώς αποκρισταλώνονται. Και στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με την Κεντρική Αφρική συνολικά θα υπογράψει το Καμερούν τη συμφωνία και πώς ε, θεωρείτε ότι αυτό θα πλήξει την οικονομική κατάσταση της χώρας σας. Θα με ενδιαφέρει πολύ να τα μάθω αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, Ντεβιτ Κάμπελ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Στην έκθεση του κυρίου Μάρτιν ε, την ε, λέξη συμμετρική από ό,τι έχω καταλάβει στο παρελθόν έχει ασκηθεί ιδιαίτερη κριτική από την Αφρική και από την Καραβική για τις CPAs, για τις ε, συμφωνίες ότι είναι σχεδόν νεοαπικιακές και ότι αναγκάζονται να ανοίξουν νέε αγορές στο Κανεμερούν χωρίς να δίνουν πολλά ως αντάλλαγμα. Αναρωτιόμουν αν το Καμερούν πιστεύει ότι του ασκείται υπερβολική πίεση εδώ, γιατί υπάρχει τεράστια διαφορά δύναμης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και του Γκούσας κράτους ε, και άλλα κράτη δεν έχουν υπογράψει. Βλέπετε να υπάρχουν μειονεκτήματα σε αυτή την συμφωνία σχέση, ε, γιατί εγώ δεν έχω δει πολλές τέτοιες συμφωνίες να έχουν έρθει σε αυτή την Επιτροπή. Υπάρχει υπάρχει ένα μεγάλο μειονέκτημα για εσά και είστε έτοιμοι να πληρώσετε αυτό το τίμημα για να έχετε πρόσβαση στι ευρωπαϊκέ αγορέ. Από την Κομισιόν, ποιο είναι εδώ, κύριο Τόμσον. Ναι, όπω πάντα, Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που παρευρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ. Γιατί ουσιαστικά έχουμε δώσει κάποια έγγραφα για αυτή τη συμφωνία το Δεκεμβρίου του 2012. Νομίζω ότι είναι διαθέσιμα και στα αγγλικά και στα γαλλικά, επομένως ε, δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα δελτία. Θα αναφερθώ ε, στα όσο είπε ο κύριος ε, Μάρτιν. Συμφωνούμε και νομίζω ότι και ο κύριος Πρέσβης αναφέρθηκε σε κάποια πολύ σημαντικά θέματα κατέστησε σαφέ ε, ότι χρειάζεται το Καμερούν τη συμφωνία, γιατί και αυτό μα καθησυχάζει ότι κάνουμε πράγματα που χρειάζονται οι άνθρωποι. Νομίζω ότι το θέμα που τέθηκε από πολλού ομιλητέ μόλι τώρα αφορά καταρχήν την υπογραφή και την περιφερειακή ολοκλήρωση. Καταρχήν, η υπογραφή έλαβε χώρα στι 15 Ιανουαρίου 2009. Α μιλήσουμε πια για την υπογραφή. Το θέμα τώρα είναι η εφαρμογή μη τη συμφωνία. Έχει γίνει η υπογραφή. Τότε, περιφερειακές πτυχές αυτού. Η περιφερειακή πτυχή καταρχήν είναι μια επιλογή για την περιοχή. Αν η περιφέρεια συλλογικά θέλει να προχωρήσει και υπήρχε βούληση συγκεκριμένα το 2007 να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά κατόπιν ε, ε, εξαφανίστηκε κατά κάποιο τρόπο το 2007. Τότε το Καμερούν είπε θέλουμε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία και θέλουμε να την αποκαλέσουμε μια συμφωνία για την Κεντρική Αφρική για να αφήσουμε την πόρτα ανοιχτή, έτσι ώστε και οι φίλοι μας από την Κεντρική να μπορούν να ενταχθούν αργότερα αν το επιθυμούν. Αυτό δεν εμποδίζει την περαιτέρω διαπραγματεύσεις να συνεχιστούν σε καθολικό περιφερειακό επίπεδο και έχουν συνεχιστεί ε, με έναν ε, τρόπο ε, που είχε την εξή συνέπεια. Οι επίσημε διαπραγματεύσει αποσυρθήκαν και είχαμε μόνο άτυπες επαφέ. Έχουμε συναντήσει τον νέο επικεφαλή αυτή την εβδομάδα, τον επικεφαλή της ΕΚΑΣ που είναι η άλλη περιφερειακή οργάνωση. Ε, και οι δύο φαίνεται να είναι ρεαλιστές και τώρα περιμένουν ε, την εντολή από το Υπουργείο για να ξαναρχίσουν οι περιφερειακές διαπραγματεύσεις. Εμείς από την πλευρά μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γι' αυτό από την πλευρά της κοινότητας ε, και της Κομισιόν από την 1η Ιανουαρίου 2008 εφαρμόζουμε τη συμφωνία και είναι δύσκολο να είμαστε πιο ευέλικτοι για την πρόσβαση στις αγορές, την πρόσβαση χωρίς δεσμούς. αναφερθήκε συμμετρία, συνοδευτικά μέτρα υλοποιήθηκαν και ήμασταν ευέλικτοι έχουν βέβαια από τότε γίνει και κάποιες διαπραγματεύσεις για τους κανόνες προέλευσης. Τώρα για το θέμα των εσόδων. Υπήρξαν μελέτες, δεν είμαι εμπειρογνώμονας, δεν είμαι ειδικό, αλλά υπάρχει ένα έγγραφο από τον ECTPM για την απελευθέρωση, την εμπορική απελευθέρωση ε, της φορολογικής προσαρμογής στην περίπτωση των EPA στην Αφρική. Και ξέρω ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο που το εξέτασαν ε, ε, οι φίλοι μας στο Καμερούν ε, και σωστά συνεχίζουν να πράττουν. Δεν ξέρω αν κάλυψα όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν αλλά ελπίζω αυτά τα, fact sheets να σας βοήθησαν. Και να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που αυτό το Κοινοβούλιο έχει εξετάσει αυτή τη συμφωνία. Υπήρξε ένα ψήφισμα σχετικά στις 25 Μαρτίου 2009. Αν και μόλις λάβαμε την επίσημη ανακοίνωση από το Συμβούλιο, εγώ αυτό μπορώ να σας πω ότι το Κοινοβούλιο έχει εξετάσει το θέμα αυτής της συμφωνίας και μάλιστα διαθέτησε και ψήφισμα το Μάρτιο του 9. Πρόεδρος, έχετε κάποια απάντηση, γιατί χρειάστηκε τόσα χρόνια το Συμβούλιο να στείλει τη συμφωνία αυτή στο Κοινοβούλιο γλώσσες. Μάλιστα. Δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ τις διευμηνείς που θα μας ε, δώσουν ακόμα 10 λεπτά. Και ας ξαναδώσουμε το λόγο στον πρέσβη του Καμερούν, γιατί τέθηκαν ε, πολλές ερωτήσεις ε, σε αυτόν. Τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σαφής. Αν δεν ήταν ενδιαφέρουσα αυτή η συμφωνία για μας, μα δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ. Το είπα και το ξαναείπα. Τη χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία, τι θέλουμε. Γι' αυτό και επέμεινα ότι σε μια διαπραγμάτευση χρειάζονται υποχωρήσεις και από τις δύο πλευρές. Κύριε Τόμψον, έχετε δίκιο, αλλά το θέμα της ευελιξίας είναι κάτι που θα πρέπει να το ξαναδούμε. Τι είναι ευελιξία? Και θα πω εδώ ότι αυτό που ζητάμε και απευθύνομαι στην Επιτροπή είναι να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Ας αναρωτηθείτε γιατί υπάρχει αδιέξοδο σε όλα αυτά τα σημεία των διαπραγματεύσεων. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για αυτοκτονία για μας. Και εμείς και οι άλλες χώρες θέλουμε αυτήν την συμφωνία. Την χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε καλύτερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές. Έχουμε πολλά χρόνια εμπορικές σχέσεις με την ε, Ευρώπη. Αλλά για να γίνει αυτή η συμφωνία πρέπει να υπάρξει προηγουμένως περιφερειακή συμφωνία. Μας λέτε ότι σαφώς στηρίζεται και τα συμφέροντα των άλλων χωρών, των άλλων εταίρων. Σε αυτή την περίπτωση λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις. Εγώ δεν μπορώ σήμερα να εκτιμήσω τις αρνητικές συνέπειες, αλλά σας ζητώ να λάβετε υπόψη σας τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει. Επαναλαμβάνω ότι δεν θέλουμε να διακοπεί η συμφωνία. Και από την αρχή είπαμε και επαναλάβαμε, το ξέρει η Επιτροπή, δεν ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη, αλλά λάβαμε υπόψη μας μόνο το εμπορικό κομμάτι. Και σήμερα έχουν προσθεθεί κάποιες επιπλέον πτυχές, αλλά αυτό που λέμε και επαναλαμβάνω θέλουμε τη συμφωνία, απλώς θέλουμε να συμπεριληφθούν και κάποια άλλα στοιχεία. Πρόκειται για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και ελπίζω την επόμενη φορά να είναι από μέρους του Καμερούν ειδικοί που να μπορούν να μπουν στην ουσία της συμφωνίας. Επαναλαμβάνω όμως, σαν γενική παρατήρηση, ναι στη συμφωνία και ναι σε περισσότερη ευελιξία και για μας και για τους εταίρους μας από την Ευρώπη. Θέλουμε να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και εμείς στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές και γι' αυτό και είμαστε υπέρ αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Είσαστε σαφείς, σαφέστατος, θέλετε τη συμφωνία, επιθυμείτε τη συμφωνία. Ο Ντέιβιτ Μάρκινγκ για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι εξίσου σύντομος. Καταρχάς δεν τίθεται θέμα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα για το ότι το Καμερούν θα υπέγραψε τη συμφωνία μόνο για εκείνο και αυτό έχει δημιουργήσει κάποιε εντάσεις ανάμεσα στο Καμερούν και στου γείτονέ του. Όμω είναι απόλυτα λογικό για το Καμερούν να υπογράψει ε, αυτή την σύμφωνη προστασία του εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζουμε και οι υπόλοιπε κεντροαφρικανικέ χώρε να επανεκκινήσουν τι ε, διαπραγματεύσεις για το εμπόριο. Η Γκαμπόν βρίσκεται σε πολύ ενδιαφέρουσα θέση, διότι δεν υπάρχουν κάποιες ε, ξεκαθαρές θέσεις τους από το 2014 βέβαια και μετά που θα ισχύσει το νέο, η νέα συμφωνία σύνδεσης θα αποτελέσει ενδεχομένως ένα κίνητρο για εκείνους να επιθυμήσουν να συνεργαστούν. Από, για τις άλλες πέντε τώρα χώρες της περιοχής αυτής υπάρχουν λιγότερα κίνητρα. Όμως ε, αυτό δεν αφορά μόνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφορά και την Κεντρική Αφρική ως περιοχή. Είναι μια πολύ αδύναμη περιοχή από πλευράς ολοκλήρωσης, ακόμα και για αφρικανικά πρότυπα. Εμείς έχουμε αυτόν τον στόχο και τον έχουμε πάρα πολύ καιρό να βελτιώσουμε την ε, ολοκλήρωση της περιοχής αυτής. Ο πρέσβης δεν ήταν τόσο ξεκάθαρος όταν μίλησε για ευελιξία, όμως μπορούμε να βοηθήσουμε στην βελτίωση της ε, ικανότητας ε, των ε, κεντρικοαφρικανικών αυτών χωρών να εισέλθουν πάλι σε διαπραγματεύσεις μαζί μας και ελπίζω να διευκολύνει την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στο στάδιο όμω που είμαστε, προτείνω να υποστηρίξουμε αυτήν την ενδιάμεση συμφωνία και όπως είπε και ο κύριος Τόμσον, ήδη την έχουμε εγκρίνει με προηγούμενο ψήφισμα, ήδη την έχουμε χαιρετήσει. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ολοκληρώνει τις ε, συζητήσεις μας. Ε, τώρα Στην επόμενη συνεδρίασή μας το Μάρτιο θα εξετάσουμε τις επιμερούς λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Να σας προειδοποιήσω ότι αύριο υπάρχει γενική απεργία στις Βρυξέλλες. Εμείς πρέπει να είμαστε εδώ στις 9 το πρωί. Για να ακούσουμε τον Επίτροπο Ντεγκούχτ. Ευχαριστώ.